Äh, Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι που είστε πάλι εδώ Ξαναρχίζουμε με τη συνεδρίασή μα. Ξεκινήσουμε τη γερμανική ώρα δηλαδή. 3 παρα 25. Χαίρομαι για το γεγονό ε, που έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, της ε, στρατηγικής εμπόριο για όλους, trade for all. Και κατά συνέπεια οι φοιτητές και οι φοιτήτριε ε, που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα διεθνού εμπορικής πολιτικής από το Παρίσι θα μας παρακολουθήσουν σήμερα εδώ. Του καλωσορίζω λοιπόν θερμά. Γιατί πράγματι οι παράμετροι του εμπορίου το ε, τελευταίο έτος μεταβλήθηκαν αρκετά. Καταρχήν δεν συζητούμε πλέον τη συμφωνία TTIP. Αλλά έχουμε πολλές διαμάχες με ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα το, τις ορμόνες στο κρέας, με το χάλιβα, τις ελιές και ένα, ζητώ, ένα, ένα σώρο άλλα ζητήματα συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΠΟΕ. Δηλαδή η συνεργασία μας δεν είναι εκείνη που αναμέναμε στο παρελθόν. Επίσης, υπάρχει μια όλο και πιο κριτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση ε, στην κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Και τίθεται δηλαδή το ερώτημα του ποιο είναι ο αντίκτυπο, ποιε είναι οι συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση και κατά πόσο ε, η υπόσχεση τη παγκοσμιοποίηση ω προ την αύξηση τη ευημερία για όλου πράγματι έχει ευοδοθεί και πώ μπορεί η εμπορική πολιτική να συνεισφέρει σε αυτό. Και φυσικά έχουμε και κάποιες αξιώσεις ως προς την ε, εμπορική πολιτική η οποία έχει ε, πλέον μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τη σήμερα ημέρα κανείς δεν συζητά πλέον τους δασμούς. Αυτά που συζητάμε σήμερα είναι συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλέον η εμπορική πολιτική. Όπως και το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, για παράδειγμα την πολιτική σε σχέση με την ισότητα των φύλων την φόρο αποφυγή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και ούτω καθεξής. Μία σειρά λοιπόν από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ε, άπτονται αν θέλετε ή σχετίζονται με την εμπορική πολιτική. Και βέβαια αυτές οι αξιώσεις σχετίζονται με το ερώτημα του πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη με αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο ευσεβείς πόθους αλλά και αυτά πραγματικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν έχει μεταβληθεί το περιβάλλον άσκησης της πολιτικής μας και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξετάσουμε εάν ε, θα πρέπει να αναθεωρεί, αν θα πρέπει να μεταβληθεί η στρατηγική μας straight for all ή όχι έτσι ώστε να είναι πράγματι έτοιμη εντό εισαγωγικών για το μέλλον. Καλώς ορίζω λοιπόν εδώ θερμά και την επίτροπό μας ε, την κυρία Μάλμστρομ που περιλαμβάνεται και στο πρώτο πάνελ των ομιλητών. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Ρέωτιγκ, τον Περιφερειακό Γραμματέα της Uni Europa, τον κύριο Αμπρουτσίνη, τον επικεφαλή εκτελεστικό διευθυντή της Eurochambers και καλωσορίζω την κυρία Κάμετς, καθηγήτρια του Bristol Law School. Ένα λοιπόν πάνελ με διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι θα αναφερθούν σε αυτό το ζήτημα και καθώς ε, εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς τους ομιλητές και απλώς έκανα την παρουσίαση εδώ, δίνω απευθείας το λόγο στην επιτροπή την κυρία Σεσίλα Μάλμστρομ. Πρόεδρε, αγαπητοί, αγαπητά μέλη του πάνελ, αγαπητοί ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι, ε, νομίζω είναι και η ώρα για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, μιλήσατε επιγραμματικά για πολλά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για το μέλλον και πρέπει να συζητήσουμε. Θα ήθελα να κάνω μια γενική επισκόπηση για το τι έχει συμβεί από την τελευταία φορά που παρουσιάσαμε την Συμφωνία Εμπόριο για Όλους και που αποτελεί και τη βάση συζήτησης. Φυσικά μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πλαίσιο, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί. Καλό είναι να κάνουμε και τη σημερινή συζήτηση για να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Θα ακούσω με μεγάλη προσοχή και του ομιλητές του πάνελ ε, και εσάς, ε, γιατί έχουμε και μια εμπορική πολιτική που θα αναγγείλουμε σε καμιά δύο εβδομάδες στην πολιτική. Θέλουμε να αξιολογήσουμε, να καταγράψουμε το που έχουμε φτάσει. Αν όχι να, κάνουμε μια, να βάλουμε μια τελεία, αλλά να σκεφτούμε που φτάσαμε και να δούμε ότι αυτή η, πολιτική, η εμπορική πολιτική δεν έχει αποκλεισμού. Γενικά τα πράγματα στην Ευρώπη πηγαίνουν καλύτερα, θα έλεγα. Ε, μειώνεται η ανεργία. Έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με άλλους, έδειξε ότι είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις. Έχουμε χώρες, ε, τρίτες χώρες που έρχονται προς εμάς και μας λένε ότι θέλουν να κάνουν εμπόριο μαζί μας. Και αυτό είναι θετικό. Φυσικά έχουμε πολλά προβλήματα. Και δεν πρέπει να επαναπαυτούμε τώρα. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα που το φίξατε ότι πολλοί πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αισθάνονται ότι το εμπόριο είναι κάτι που του αφορά ή φέρνει καρπού για αυτού. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο είναι για όλου. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο τη δουλειά που κάνουμε με αυτή την ανακοίνωση εμπόριο για όλου. Θέσαμε το όραμα πριν από δύο χρόνια. Το όραμα δηλαδή είναι να εξασφαλίσουμε ότι η εμπορική πολιτική δίνει πράγματα απτά στου Ευρωπαίου πολίτε. Είναι λειτουργική για του εργαζόμενου, για τι εταιρείε και του καταναλωτέ επίση. Μετά από δύο χρόνια είναι πολύ σωστό να κάνουμε μια αποτίμηση του πού έχουμε φτάσει. Θα σας πω τι ξέρουμε και θέλω να ακούσω τις δικές απόψεις για αυτά. Για το, το πώς θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτή τη φιλόδοξη ατζέντα, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις αξίες μας, ούτως ώστε να υπάρχουν πρότυπα για περιβαλλοντικά θέματα, εργατισιακά θέματα και στην Ευρώπη, αλλά να τα προωθήσουμε και στους εταίρους μας. Πώς θα αυξήσουμε τη διαφάνεια και πώς η μεγαλύτερη διαφάνεια θα αυξήσει την εμπιστοσύνη και την καλή συζήτηση, την επικοδομητική συζήτηση. Έχουμε μια πολιτική για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Εσείς που είστε εκπρόσωποι των διαφόρων ε, ενδιαφερομένων φορέων θα μας κατευθύνετε στις προτάσεις μας. Λοιπόν, ποια είναι η πρόοδος που έχουμε ε, σημειώσει και τα, ποια είναι τα κενά. Καταρχάς, θέλουμε μια εμπορική πολιτική που να είναι αποτελεσματική. Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά πραγματικά τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε. Ε, έχουμε το εμπόριο στις υπηρεσίες. Ε, οι υπηρεσίες είναι και πιο σημαντικές. Κανονιστική συνεργασία για να προστατεύουμε τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό εδώ. Εδώ το έχουμε προχωρήσει, προωθήσει και με τον Καναδά και με την ε, Ιαπωνία. Επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό εμπόριο σε διάφορες διαπραγματεύσεις και στον ΠΟΕ και το σπρώχνουμε και στην ε, ε, Υπουργική στον Πουένος σε λίγες εβδομάδες. Ε, επίσης στην εφαρμογή εστιάζουμε και θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο ε, κάνουμε μια επισκόπηση του, του που έχουμε φτάσει στις εμπορικές μας συμφωνίες και μια ε, ε, πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε λέει ότι υπάρχουν απτά αποτελέσματα των εμπορικών συμφωνιών με αύξηση των εξαγωγών, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να αδράξουμε όλες τις ευκαιρίες. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε μαζί σας στο Κοινοβούλιο, αλλά και, σε εταιρική, και είσαστε εταίροι μα για την εφαρμογή. Υπάρχουν ειδικέ διατάξει για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει, ώστε να τι ε, ενθαρρύνουμε να υποφεληθούν από τι ε, συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Έχουμε ειδικό κεφαλαίο τη μικρομεσαίε στην συμφωνία με την Ιαπωνία. Και ελπίζουμε ότι την έχουμε και σε άλλε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν όλα αυτά και ότι το εμπόριο είναι υποφελέ. Για να είναι υποφελέ θα πρέπει να είναι δίκαιο. Θα πρέπει όλοι να παίζουν με του κανόνε. Γι' αυτό ε, δεν θέλουμε διακριτικές μεταχειρήσεις κατά των Ευρωπαίων ε, επιχειρήσεων με όλα τα μέσα και μέσω του ΠΟΕ, ε, μέσω του Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ, αλλά και μέσω των εργαλείων ε, ε εμπορικής άμυνας. Το 2016 έχουμε λύσει 20 υποθέσεις ε, που αφορούν 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγών. Πολλά λεφτά είναι αυτά εξυγχρονίζουμε τα ε, εργαλεία εμπορικής άμυνας και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω μέχρι το τέλος του 2017 να είμαστε σε θέση να πούμε ότι τα έχουμε καταφέρει 100% εκεί. Πάμε στο δεύτερο πυλώνα, αξίες. Σημαίνει καταρχάς πάνω απ' όλα ότι καμιά ευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία δεν θα μειώνει τα δικά μα πρότυπα για το περιβάλλον, για τα εργασιακά, για του καταναλωτέ ή την κοινωνική προστασία. Είναι οι Ευρωπαίοι νομοθέτε που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα και όχι οι εμπορικέ συμφωνίε. Επίση, προωθούμε αυτά τα πρότυπα στο περιβάλλον. Στην Ιαπωνία στην ε, συμφωνία με την Ιαπωνία για πρώτη φορά ρητά ε, αναφερόμαστε και υποστηρίζουμε την ε, Συμφωνία των Παρισίων και θα γίνει και στις μελλοντικές συμφωνίες το ίδιο. Επίσης, ε, έχουμε διάταξη ε, βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις συμφωνίες. Η ανάπτυξη αυτή ε, είναι στην καρδιά και των μονομερών προτιμησιακών συστημάτων και των γενικευμένων προτιμήσεων πλάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δράει εκεί που υπάρχουν ανησυχίε και έχουμε σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη γιατί όπως ξέρετε συζητάμε μαζί σας και με πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για το πώς θα ενισχύσουμε την, το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης και το θέμα της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Κοιτάμε το πώς οι εμπορικές πολιτικές μπορεί να βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, να προωθήσουμε και θα έχουμε ένα κεφάλαιο στην συμφωνία με το Μεξικό για πρώτη φορά ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε το δίκαιο και δεντολογικό εμπόριο και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις ε, γυναίκες στο εμπόριο. Πρόσφατα ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τη Χιλή και για πρώτη φορά θα έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο για τις ε, γυναίκες και το φύλλο, τη διάσταση του φύλου και περιμένω με υπομονησία τα σχετικά αποτελέσματα. Επίσης έχουμε μαζί με εσά πετύχει ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, ο καονισμός για τα μεταλλεύματα, ε, τα ορυκτά μεταλλεύματα όπως το τανξτένιο κτλ. Και έχουμε απαγόρευση αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούν για βασανιστήρια ή θαντική ποινή. Και έχουμε μια παγκόσμια συμμαχία στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο με 58 χώρες σε όλο τον κόσμο και περισσότερες που θα ενταχθούν στο μέλλον. Επίσης, Έχουμε κάνει πολλά σε ό,τι αφορά το εμπόριο με πιο διαφανή τρόπο και είμαι περήφανη για τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει. Ήσασταν πολύ υποστηρικτικοί, σας ευχαριστώ γι' αυτό, ούτως ώστε οι εμπορικές διαπραγματεύσεις να είναι πιο διαφανείς. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, εμείς είμαστε πρωτοπόροι εδώ, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Δημοσιεύουμε όλα τα κείμενα για τις νέες διαπραγματεύσεις, για τους γύρους, ε, επεξηγηματικό υλικό και όλα αυτά είναι σε μία ενία επιγραμμική πλατφόρμα με πληροφορίες για, τα, για τις έρευνες, για το εμπόριο κτλ. Όλες τις πληροφορίες είναι εκεί. Συστηματικά, και το κάνετε κι εσείς, ζητάμε από το Συμβούλιο να δημοσιεύει τις διαπραγματευτικές εντολές. Έγινε στο TTIP με τη ΣΕΤΑ και με την TISA και πρόσφατα με την Επονία. Ε, αποφασίσαμε για πρώτη φορά να δημοσιεύσουμε ένα σχέδιο ε, διαπραγματευτικής οδηγίας για την συμφωνία με την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Σας τη στείλαμε απευθεία, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια, ούτως ώστε να ξεκινήσουν την δουλειά πάνω σε αυτά. Ίσως όταν το Συμβούλιο τα, τα υιοθετήσει αυτά κείμενα, αλλάξουν λιγάκι. Αλλά ο σκελετό θα είναι αυτός, ούτως ώστε θα μπορείτε να ξέρετε εκ των προτέρων περί τίνος πρόκειται ούτως ώστε οι διάφορες επιτροπές να αρχίσουν την, να, κινούνται και να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Είναι ένα βήμα αυτό που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη, πιστεύουμε, και θα μειωθούν οι μύθοι που υπάρχουν για την εμπορική πολιτική. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί και η νομιμότητα της διαδικασίας. Επίσης, κάθε μέγιστη, κάθε μείζωνα πρωτοβουλία που προωθούμε, τη βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση και έχουμε πολλές δημοσίες εκδηλώσεις όπου καλούμε οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών για να συνεισφέρουν. Έχουμε αυτή τη μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή με την κοινωνία των πολιτών που μπορεί να μας συμβουλεύσει για όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να μας ε, βοηθήσει με τις γνώσεις της στη διαπραγμάτευση. Έχουμε μεταρρυθμίσει το ISDS, δηλαδή τη διαβόητο, το διαβόητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών ε, κράτους ε, επενδυτών με μεγάλη δημόσια διαβούλευση, τα τη θυμάστε. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση τώρα που έχουμε απέναντι στον Καναδά, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Πιο διαφανή, πιο προβλέψιμη στάση και θέλουμε να κάνουμε ένα ε, πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο μαζί με, άλλους, μαζί με άλλες χώρες κάνουμε προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλες αυτές τις αρχές τις προωθούμε και σε δημόσιο επίπεδο και σε περιφερειακό και σε πολυμερές. Φυσικά ο κρυγονίας λίθος είναι ο ΠΟΕ, ε, η συμφωνία για τις ε, πληροφορίες τις τεχνολογικές, ε, η συμφωνία για την διευκόνιση του εμπορίου πέστη πολύ σημαντική. Έχουμε μια έκθεση για την εφαρμογή του εμπορίου για όλους πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος Γιούνκερ τον ανέφερε, την ανέφερε στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και μπορείτε να διαβάσετε σε αυτήν την ομιλία περισσότερες λεπτομέρειες. Η, ε, συμφωνία με τον Καναδά μπήκε σε εφαρμογή και αρχίσαμε διαπραγματεύσει με πολλές άλλες χώρες για το θέμα αυτό. Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν. Πάρα πολλά έχουν γίνει. Φυσικά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Περιμένω τη σκέψη σας για το τι μπορεί να βελτιωθεί, γιατί φυσικά το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός συνεισφέρει στην σε μια ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη. Πρέπει όμως να συμπληρωθεί μέσω ενεργών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο κυρίως, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο εμπόριο, ούτως ώστε οι επιπτώσεις ε, της παγκοσμιοποίησης να είναι δίκαιες και προστατεύουν τις αξίες μας και βασίζονται σε ένα σύστημα με κανόνες. Έτσι, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ε, επωφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση, αλλά και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή της. Μια πολιτική που θα προωθεί τις αξίες εντός και εκτός, ε, έχει, θέτει ψηλά πρότυπα και στρέφεται σε φίλους και συμμάχους ε, σε όλο τον κόσμο για να προωθηθούν αυτές οι βασικές αξίες. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε με την παγκόσμια διακυβέρνηση, θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, προσπαθούμε να το κάνουμε μέσω πολλών ε, διμερών ε, δράσεων, να δημιουργήσουμε ένα κύκλο φίλων για να έχουμε ένα παγκόσμιο ανοιχτό εμπόριο. Το εμπόριο είναι καλό για την οικονομία, αλλά πρέπει φυσικά να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες και εμείς και μαζί με άλλους εταίρους, ούτως ώστε να έχει πρακτικά αποτελέσματα στον κάθε πολίτη. Εδώ φτάσαμε και προσβλέπω σε μια εποφελή συνεργασία. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε και αυτό το πάνελ. Ευχαριστούμε, Σεσίλια. Comprehensive Yeah, It's working. Before giving the floor to panelists, Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ομιλία. Πρωτού δώσω το λόγο στους επόμενους πάνελες, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας σε ό,τι αφορά την έκθεση εφαρμογής ε, της κοινής ε, πολιτικής. Ε, πολιτικής, η κυρία Σαϊφ, Λοιπόν, να πω φυσικά ότι πρόκειται για μια συνεδρίαση με web streaming. Οπότε, οι τηλεθεατές μας μέσω του ίντερνετ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα μέσω Twitter. Στο hashtag Trade Policy Day. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή διεύθυνση για την υποβολή των ερωτημάτων μέσω Twitter. Ακούσαμε λοιπόν την συνοπτική έκθεση στο προς το που βρισκόμαστε Αλλά τώρα να περάσουμε στον κύριο Ρότινγκ, ο οποίος εκπροσωπεί γύρω, στους 20, ε, γύρω εκατομμύρια εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών. Ε, τι νομίζετε λοιπόν ως προς το Πού βρισκόμαστε από οικονομική άποψη και σχέση με την εμπορική πολιτική. Φυσικά βρίσκομαι εδώ πρώτα απ' όλα ως ε, Γενικός Γραμματέας της Uni Europa, αλλά ε, εκπροσωπώ και έναν άλλο διεθνή οργανισμό εκπροσωπούμε 20 εκατομμύρια εργαζομένους ε, σχεδόν σε όλες τις χώρες όπου επιτρέπονται τα συνδικάτα. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, εμάς η ανησυχία μας είναι οι επιχειρήσεις και κυρίως οι εργαζόμενοι. Χάρη σε αυτούς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο είναι καλό να αναφερθούμε και στην εκδήλωση της προηγούμενης εβδομάδας ε, στο Γκέτενμπορ και το ε, πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αλλά είναι καλό να ε, επηρεάζει και την προσέγγιση των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο. Από την άποψη ενός συνδικάτου οι εμπορικές συμφωνίες και οι εμπορικές συναλλαγές είναι, πρέπει να βελτιώσουν ε, τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Σημασία δεν έχει μόνο το κέρδος και η οικονομία. Πρέπει να επωφεληθεί και ο πληθυσμός. Θέλουμε μια βιώσιμη, δίκαιη και κοινωνική προσέγγιση που διαφαλίζει φυσικά την ανταγωνιστικότητα με βάση φυσικά την ποιότητα και όχι το dumping. Και αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, το ε, ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι κάτι που μπορούμε να εξάγουμε. Και όπως είπε η κυρία Επίτροπος, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα του εμπορίου ε, επηρεάζουν την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι συνδικάτων, πρέπει να βλέπουμε την εμπορική πολιτική ως μέσο για να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων ε, είτε από ε, δημόσιες, ε, είτε από ιδιωτικές εταιρείε, είτε από κυβερνήσεις στις χώρες με τις οποίες συναλλασσόμαστε πριν από ε, χρόνια είχαμε ε, μια υπόθεση με μια ισπανική εταιρεία στην ε, Νότια Αμερική, στην οποία είχαν παρατηρηθεί κάποιες παραβιάσεις. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορικές συναλλαγές και οι συμφωνίες μας δεν παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα όταν ε, εξετάζουμε το τομέα των υπηρεσιών μεταξύ άλλων πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ε, ε, φυσικά Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για άλλες χώρες του κόσμου. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, οι εμπορικές συμφωνίες ε, πρέπει να προσπαθούν να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Και θα μπορούσαμε να ε, συμφωνήσουμε σε ένα κεφάλαιο σχετικό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στις εμπορικές συμφωνίες. Είναι σημαντικό να προβλέπονται οι απαραίτητες ε, διασφαλίσεις και εγγύησεις. Υπάρχουν μηχανισμοί ε, ε, κρατικοί, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμβάλλουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι τα πρότυπα και οι συμβάσεις πρέπει να τηρηθούν, αλλά πρέπει να στρέψουμε και το βλέμμα μας παραπέρα. Πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι ε, αξιοπρεπείς αποδοχές. Κάποιοι θα θυμούνται ε, το ατύχημα στο Ράνα Πλάζα του Μπαγκλεντές όπου οι συνθήκες εργασίας ήταν τόσο άσχημες ε, που πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. τα συνδικάτα και η κοινωνία των ε, πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και είναι το ίδιο σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των συμφωνιών η κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι να συνεισφέρουν. Γιατί δεν ε, αναπτύσσουμε έναν ε, συνολικό κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας. κυρίως όταν κοιτάμε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Νότια Αμερική και στην Ιαπωνία, οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να συνδέονται στενά με την εμπορική πολιτική προκειμένου να διασφαλίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ε, συνεισφορά των εργοδοτών στις σχετικές συζητήσεις. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλη την αλυσίδα αξίας και όταν υπάρχει καλός κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη, αυτό είναι θετικό, αλλά δεν βοηθάει όταν έχουμε ε, μία σειρά επιχειρήσεων σε όλο το κόσμο. Σας προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική πολιτική και τη Συμφωνία της Ελεύθερων Συναλλαγών για να προωθήσουμε την πολιτική μας σε όλο τον κόσμο, να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχουν, μιας και υπάρχουν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, γιατί να μην διευρύνουμε ε, αυτό το θεσμό και ε, σε όλη την παγκόσμια λυσίδα αξιών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής μας. Το δεύτερο σημείο είναι οι γενικές ανησυχίες των συνδικάτων και σε πρώτη ε, κυρίως ό,τι αφορά το σύστημα επίλυσης διαφορών, αυτό το σύστημα θα επιφέρει βελτιώσεις, δεν είμαστε όμως ακόμα υπέρ και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν τα συστήματα που ε, υπάρχουν ήδη και προβλέπονται σε κάθε χώρα για την αντιμετώπιση ε, αιτιάσεων. Θυμάμαι, ε, έχω διαβάσει για το σύστημα που υπήρχε στο, το 19ο αιώνα ε, στην ε, Κίνα, όπου ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε όλοι να τηρούν τα, τις νομικές διατάξεις μας, πρέπει να προβλέπονται τα σχετικά πρότυπα και όσοι υπογράφουν ε, τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να τηρούν όλες ε, τις ε, διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τη ρυθμιστική συνεκτικότητα ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των εθνικών κοινοβουλίων. Και κάποιες φορές έχουμε αμφιβολίες όταν Ξετάζουμε κάποιες ε, προτάσεις, όχι απαραίτητα της Κομισιόν. Και ε, επανέρχομαι στη διάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων για να προχωρήσουμε. Καλό θα ήταν το Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ε, αναπτύξουν ένα κεφάλαιο που αφορά τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους και όταν κοιτάμε όλους τους ε, τομείς και κυρίως τους εγκάρσιους τομείς ε, στην Ευρώπη, θα ήταν καλό να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ένα σαφές ε, μήνυμα από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όταν εγώ συζητώ την εμπορική πολιτική, συχνά ακούω την άποψη ότι ε, το εμπόριο τελικά αποβαίνει προς, στο προς όφελος αν δείτε, των ε, πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ε, κυρία Μπρουτσίνη, από την πλευρά των Euro Chambers, ποια είναι η δική σας άποψη σε με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πραγματικότητα το εμπόριο δεν ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις. Ε, ευνοεί και αποβαίνει προς όφελος του ε, συνόλου της κοινωνίας, των πολιτών και όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, ε, στην αλυσίδα ε, των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Και θα ήθελα να επιμείνω λίγο εδώ στην πλευρά των επιχειρήσεων. Όταν αγοράζουμε ή ε, πουλάμε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία στην αλλοδαπή, το κάνουμε γιατί υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να το πράξουμε. Δηλαδή, επειδή είναι ένα καλύτερο προϊόν ή έχει μια ευνοϊκότερη τιμή ή πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο δεν υφίσταται εκεί όπου ε, βρισκόμαστε. Δηλαδή το εμπόριο είναι πολύ ξεκάθαρο προς το στόχο του. Προσπαθεί κανείς να εξασφαλίσει κάτι το οποίο είναι ή καλύτερης ποιότητας, είναι ευθυνότερο ή δεν είναι διαθέσιμο κάπου. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση, τότε πολλά από τα όσα αναφέρθηκαν και τα οποία εκτιμώ, δεν ανήκουν αμυγός στον, σε αυτό το τομέα της, του εμπορίου. Αφορούν δηλαδή την κοινωνία και αφορούν γενικότερα τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε, αλλά όχι συγκεκριμένα το εμπόριο. Δεν αφορούν συγκεκριμένα το εμπόριο. Και αυτό το λέω γιατί δεν θεωρώ ότι το εμπόριο από μόνο του μπορεί να επιλύσει όλα τα ε, προβλήματα. Αποτελεί ένα εργαλείο. Αποτελεί το ίδιο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε όταν, για παράδειγμα, διαθέτουμε στην δική μας την μεταπέα αγορά αγαθά και υπηρεσίες. Απλώς το κάνουμε σε άλλες χώρες, στην Αρδαπή. Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ότι ζητήματα ε, πολιτικής ε, δεν είναι τόσο περίπλοκα έτσι ώστε να μπορούν να επιληθούν μέσω μιας εμπορικής πολιτικής και χωρίς να χρειάζεται να περιληφθούν εδώ και άλλοι τομείς πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ε, εμπορική πολιτική η οποία θα σέβεται ε, τις προσδοκίες, το όραμα, τις προθέσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά την προσέγγιση του στην παγκόσμια αγορά. Σίγουρα θα θέλαμε εδώ να συμβούν πολλά περισσότερα. Για παράδειγμα, οι διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται ε, έχουν ολοκληρωθεί και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, στη τέληση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του να καταστεί πραγματικά παγκόσμια εμπορική μας ε, πολιτική. Θα θέλαμε να υπάρχει λοιπόν ένα παγκόσμιο πρότυπο, να υπάρχει μια παγκόσμια αγορά χωρίς εμπόδια. Κάτι τέτοιο θα το θέλαμε εμεί από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί πράγματι θα έπρεπε να όφελο των επιχειρήσεών μα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ακριβώ να ανταποκριθούμε καλύτερα στι ανάγκε των καταναλωτών. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτή την ε, πολιτική, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί ακολουθούν τις εξελίξεις τα δεκτενόμενα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα σε δύο στοιχεία, που είναι το σκέλος των υπηρεσιών, το οποίο λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, αλλά και η διάσταση της ψηφιοποίησης της οικονομίας μας. Δηλαδή, όσο περισσότερους κανόνες μπορούμε να θεσπίσουμε οι οποίοι θα διευκρινίζουμε εύκολο και σαν τρόπο αυτά τα στοιχεία, τη ρύθμιση αυτών των στοιχείων στην εμπορική μας πολιτική, τόσο περισσότερο θα ευνοηθούμε όλοι μας. Και εδώ αναφερόμενο στο Ποιο είναι τελικά ο αποφελούμενος, νομίζω πως δεν θα αποτελέσει έκπληξη για την κυρία ότι κατά τη δική μας άποψη ένα τμήμα του οικονομικού μας ιστού, αν θέλετε, το οποίο δεν έχει λάβει την απαραίτητη σημασία, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες οι οποίες απασχολούν στον εξαγωγικό τομέα, δηλαδή στα προϊόντα ε, και τις υπηρεσίες, 6 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ το 1 τρίτο των ε, ε, προϊόντων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κόσμο ε, προέρχονται από την εμπορική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρί να αναφέρουμε καν σε εκείνε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε εμπλέκονται και συνεισφέρουν στην αλυσίδα παραγωγή αξία των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει χρήζουν ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο αυτή τη πολιτική. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβούν σε εξαγωγέ κάποια στιγμή. Όχι. Ένα κλάσμα, ένα μέρος αυτών των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να εξάγει απευθεία στι διεθνεί αγορέ, αλλά για να είναι σε θέση να το επιτύχει, χρειάζεται συγκεκριμένα στοιχεία. Και τέσσερα συγκεκριμένα στοιχεία θα ήθελα να σα αφαίρω εδώ, τα οποία ε, τα μέλη μα μας αναφέρουν ότι πράγματι θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Καταρχήν, οι κανόνε σε ό,τι αφορά την προέλευση των προϊόντων. Δεν μπορώ να αναφέρω ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ο οποίο προσέρχεται στο δικό μας ε, μελτήριο, το οποίο εκδίδει και όλα τα, αυτά τα πιστοποιητικά προέλευσης και μας λένε λοιπόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν ένα τέτοιο ε, πιστοποιητικό προτιμησιακής μεταχείρισης γιατί είναι τόσο περίπλοκοι οι κανόνες. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση όλα όσα προσπαθείτε να κάνετε στο πλαίσιο της σε σχέση με τους κανόνες που θα ισχύσουν δεν θα μας ωφελήσουν σε τίποτα. Εάν πράγματι λοιπόν θέλουμε να δώσουμε περισσότερη αξία στον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τότε θα πρέπει να απλουστεύσουμε περισσότερο την προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά ε, τους κανόνες σε σχέση με την πρόληψη. Και θα πρέπει να υπάρξει ένα εύκολο στην εφαρμογή του εργαλείου. Και εδώ, όπως θα θυμόσαστε, ε, κυρία Επίτροπη, έχουμε ε, προτείνει εδώ και κάποιο καιρό μία μέθοδο υπολογισμού ε, αυτών των ε, κανόνων για την προέλευση. Αλλά θα πρέπει να είναι εύκολο λοιπόν, εύκολος αυτός ο υπολογιστή στην εφαρμογή του ε, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσει. Μία λοιπόν τέτοια μέθοδο υπολογισμού θα, ήταν, θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή αυτών των επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο τώρα στοιχείο, το οποίο ήδη αναφέρθηκε, είναι η εφαρμογή στην πράξη. Είναι πολύ καλή και επιχαίρουμε για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται τώρα να ε, παρουσιάσει μια έκθεση εφαρμογή ε, και έναν ε, χάρτη πορεία, αλλά αυτός ο χάρτης πορεία εφαρμογής αφορά τις τρίτε χώρε, αφορά τους εταίρου μας. Ενώ, από όσο εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, δεν υπάρχει ένας χάρτης πορεία εφαρμογή σε ό,τι αφορά εμά του ίδιου. Και έχουμε διαπιστώσει ότι οι τρίτες χώρες ε, αξιοποιούν πολύ περισσότερο και προωθούν πολύ περισσότερο ε, την σύναψη μια ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι εμεί. Για παράδειγμα, αν επιστρέψω στο ζήτημα των επιστοποιητικών, το περισσότερο από 90% των τρίτων χωρών, των χωρών εταίρων μας, χρησιμοποιούν αυτά τα ε, προτιμησιακά ε, πιστοποιητικά ή προτιμησιακή μεταχείριση, ενώ το ίδιο ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 70%. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, γιατί να μην υπάρξει ένα χάρτη πορεία σε ό,τι αφορά την ίδια την Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, θα ήταν περίπλοκο κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε περίπλοκοι και ω μόρφωμα, αλλά εάν μπορούμε να συντάξουμε ένα χάρτη πορεία για τι τρίτε χώρε, σίγουρα θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το να γνωρίζουμε με διαφανή τρόπο το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να κερδίσουμε από την διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με τρίτες χώρες. Τώρα, ε, το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήδη αναφερθήκατε σε αυτό, ε, κυρία Επίτροπε. Πρόκειται πράγματι για ένα σημαντικό στοιχείο. Στο πλαίσιο δηλαδή των σύγχρονων, των μοντέρων συμφωνιών που συναπούμε με χώρες. Ε, πρόκειται για ένα αμυγός ευρωπαϊκό, αν θέλετε, στοιχείο, το οποίο καταφέραμε να διαδώσουμε, αν θέλετε, και στους εταίρους μας ανά τον κόσμο, μέσω ακριβώς μιας σωστής, έστοχης διαπραγματευτικής ε, τακτικής. Και έτσι, λοιπόν, έχει καταστεί πλέον συνήθις τακτική, αν θέλετε, το να συμπεριλαμβάνεται ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Και αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί. Καταρχήν, ε, δεν αποτελεί έναν εγκάσιο αν θέλετε, κανόνα ή εγκάρσιο κεφάλαιο αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις ε, συμφωνίε, Γιατί βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τις επιπτώσεις των υπολείπων πυλώνων αυτών των, ε, των υπολείπων κεφαλών στα, στον πυλώνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής δηλαδή αντιμετωπίζεται με πιο οριζόντιο τρόπο. Και ένα τελευταίο στοιχείο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι αυτό της διαφάνειας. Σίγουρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Όχι μόνο μέσω, για παράδειγμα, τη δημοσίευση του σχεδίου ε, των εγγράφων διαπραγμάτευση, αλλά και μέσω εμπλοκή από νωρί των ενδιαφερόμενων και συναρμόδιων διαφορεών, όπω έχει συμβεί βέβαια σε κάποιε περιπτώσει, στην διαπραγματευτική διαδικασία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα ωφέλη από την στρατηγική της, του εμπορίου για όλου στο πλαίσιο τη εμπορική Η τελευταία μιλήτρια είναι από το Bristol. Είναι πρώην ε, βιομηχανικό κέντρο όπου παράγονταν αυτοκίνητα. Ακούσατε τρεις πανεβάσεις ήδη, με... Ε, όπου οι ομιλητές εκπροσωπούσαν ε, συγκεκριμένα συμφέροντα. Τώρα ποια είναι η επιστημονική άποψη για αυτή την στρατηγική εμπόριο για όλους. Καταρχάς, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ε, μεγάλη μου τιμή. Μερικά από τα αναδυόμενα θέματα που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις ε, των πανελιστών είναι η ανάγκη για διαφάνεια, βελτιωμένη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διάφορες αγορές. Εγώ θα σταθώ στις ε, κοινωνικές ε, αξίες που είναι γεγραμμένες στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το εξωτερικό, κυρίως σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες και με τον, με τον τρόπο που έχει οικοδομήσει την εμπορική της πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιφερειακός παίκτης, όχι σαν μια, ένα μπλοκ 28 χωρών, 28 χωρών, είμαστε ακόμη 28 έτσι, αλλά η Ευρώπη παίζει και ως περιφερειακός ε, παίκτη και εταίρος. Ε, προσπαθεί να επηρεάσει με τις κοινωνικές αξίες, καθολικές αξίες ε, που όπως διασφαλίζονται σε επίπεδο ΙΕ μέσω του εμπορίου. Τώρα, αυτό που άκουσα ε, είναι οι κοινωνικές αξίες και κοινωνικές αξίες για τις επιχειρήσεις μπορεί να φαίνονται ε, ασήμαντες ε, για το εμπορικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν αυτές οι εγγεγραμμένες στο άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, και επίσης και στο άρθρο 3 όπου έχουμε τις εσωτερικές μας αξίες που τις εξωτερικεύουμε μέσω των δράσεων που έχουμε σε τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμπόριο για το εμπόριο. Ε, το εμπόριο είναι ένα δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να είναι νόμιμο και εφόσον υποθέτω λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ να σκεφτούμε για να δούμε σε ποιο βαθμό το εμπόριο για όλου πετυχαίνει το στόχο του και μήπω υπάρχουν κάποιε προκλήσει και προβλήματα στην εφαρμογή του στι τρίτε χώρε ειδικά. Ξεκινήσαμε με μια συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση εδώ στο πάνελ. Η ιδέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει προς τα έξω με βάση τις δικές της αξίες. Μετά θα ακούσουμε από, το γενικό, από τον απλήρωτή διευθυντή του ΠΟΕ ε, πολλά για το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό λοιπόν. Αλλά θα πρέπει μέσα αυτήν την γενική εικόνα, σε πολυμερές πλαίσιο, να σας εξηγήσω τι κάνουμε την εμπορική πολιτική λιγάκι στα πλαίσια του εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούμε να δούμε το εμπόριο για όλους απομονωμένα. Ε, έχει φυσικά οικονομικό προσανατολισμό, αλλά παρόλα αυτά έχει και ε, εγγενείς κοινωνικές αξίες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο είναι συνεπές ως προς την αναπτυξιακή πολιτική με βάση την ατζέντα του 2030 για τις, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κτλ η δουλειά μου εστιάζεται στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με, την, ε, με τις χώρες ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για κάμια αποτίμηση για το πόσο αυτές οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου έδωσαν καρπούς, ιδίως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει, συνεχίζει τις ε, περιφερειακές εμπορικές ε, συμφωνίες ως εργαλεία ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Τα επόμενα 10 με 15 χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου ΑΕΠ θα παράγεται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. και επομένω είναι σημαντικό ε, να ε, υποφεληθούμε από αυτές τι ευκαιρίες. Μέσω των συμφωνιών αυτών έχουμε μια προοδευτική προσέγγιση. Ε, ακούσαμε σήμερα για την συνεργασία που έχουμε σε διάφορα κεφάλαια περιβάλλον, ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την καλή διακυβέρνηση, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προάγει τι αξίε τη στο εξωτερικό. Είναι επιτυχές. Αν το δείτε με τυπικούς όρους ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Όμως, το βασικό πρόβλημα που βλέπουμε με τις συμφωνίες του ελευθέρου εμπορίου είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι νομικά δεσμευτική σε πολλές περιπτώσεις. Η βιώσιμη ανάπτυξη Φερρυπίν δεν, δέχ... δεν τη δέχεται κανένα δικαστήριο ως νομική αρχή, ας πούμε, νομικά δεσμευτική. Είναι μια μήτρα ή μια αρχή όπου μέσα από την οποία προωθούνται διάφορε άλλε αξίε, όπω η ισότητα των φύλων ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα κτλ. Υπάρχουν λοιπόν διατάξει συμφωνίε ελευθερού εμπορίου μεν, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικέ αυτέ οι διατάξει. Και όπου είναι νομικά δεσμευτικέ, όπω οι καθολικέ αξίε, ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή, αν και εδώ υπάρχουν θέματα δηλαδή, και αμφισβητήσεις. Ακόμη και αν είναι ε, δεσμευτικά, δεν μπορεί κανένας να προσφύγει για τέτοια θέματα ενώπιον των δικαστηρίων. Και εκεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των, του μοντέλου των ε, Συμφωνίων Ελευθέρου Εμπορίου ανά τον κόσμο. Σήμερα άκουσα εδώ τους ομιλητές και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα εργάζονται για το καλό της παγκόσμιας οικονομίας. Το πιστεύω. Όμως, είναι σε πολύ ισχυρή θέση για να ασκήσουν την ε, πολιτική αυτή με πιο δίκαιο τρόπο. Ε, Παραδείγματο χάρη, ο μηχανισμό επίλυση διαφορών στι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Ε, στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τη συμφωνία μάλλον Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ, ε, προωθείται μέσω του πολιτικού διαλόγου και τη συνεργασία με βάση τη Συμφωνία Κοτονού και του πυλώνε για την εταιρική σχέση και τον πολιτικό διάλογο η συμφιλιωτική προσέγγιση που υπάρχει στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μοιάζει ωραία στην πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι οι εταίροι δεν είναι ισότιμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο ισχυρός εμπορικός εταίρος από τις υπόλοιπε χώρε με τις οποίες ε, διαπραγματεύεται. Αναπτυξιακά είναι πιο ισχυρή εννοώ. Σε ορισμένε περιπτώσει, σε άλλε συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου, Υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στο σύστημα του ΟΗΕ επίλυση διαφορών. Παραδείγματο χάρη η περίπτωση Ευρωπαϊκή Ένωση Περού-Κολομβία, είτε για θέματα δασμών, ε, στα αλκοολούχα ποτά. Έστω και η απειλή να προσφύγουμε αντίον τη Κολομβίας στον ΠΟΕ ήταν αρκετή για να αναθεωρηθεί η νομοθεσία τη Κολομβία και να αλλάξει κανόνε για να συμμορφωθεί με το πλαίσιο του ΠΟΕ. Αλλά αυτό είναι σχεδόν εξαίρεση στο μοντέλο των συμφωνιών Ελευθερών εμπορίου. Η προτεραιότητα είναι στις οικονομικές αξίες πάντα. Αξίες που είναι σημαντικέ είναι αυτές που έχουν σημασία για το εμπόριο και, όχι, και δεν προάγονται τόσο πολύ ε, τα κοινωνικά θέματα και το κοινό καλό, ας πούμε, που μας απασχολεί σήμερα. Η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε, Φερρυπίν, την συμφωνία ε, εμπορίου με την Σιγκαπούρη. Ε, υπάρχει πρόβλημα ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιγκαπούρη έχουν ε, τελείως διαφορετικές απόψεις για τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και όμως εδώ τα εμπορικά ε, ζητήματα είναι τα πιο σημαντικά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Από την άλλη πρέπει να σεβαστούμε και η την κυριαρχία του εταίρου μας. Ε, αν όμως συμφωνίες ελευθέρου ε, εμπορίου υπάρχουν οι κοινωνικές αξίες ε, και εφόσον το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μην στέκεται απλώς σε ρητορίες. Στι ενδιάμεσε αναθεωρήσει και σε πολλές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναγνώριση των ελλείψεων που υπάρχουν ε, σε ορισμένε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, FTAs δηλαδή. Η πενταετή αναθεώρηση των οικονομικών συμφωνιών λέει ομά ότι αυτές οι πολλές από αυτές οι συμφωνίες δεν λειτουργούν καλά. Ως ε, δικηγόρος ε, διάβασα εντυπωσιασμένη ε, με την έκθεση όπου αναγνωριζόταν ότι υπήρχαν οικονομικά ελλείμματα, ελλείμματα στην πληροφόρηση κτλ. Σε αυτή την FTA οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να καταλάβουν καν την τεκμηρίωση. Ε, πλήρωναν καλύτερα τους δασμούς για να πάρουν την προτίμηση, γιατί δεν είχαν πρόσβαση σε πληροφορίε. Ε, οι κανόνες καταγωγής είναι πάρα πολύ περίπλοκοι επίσης. Έχουμε δει ότι υπάρχει πιο πρόβλημα. Και μερικές φορέ έχουμε ε, αντικρουόμενους κανόνες καταγωγής που, καταγωγής που δημιουργεί προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αυτέ οι συμφωνίε φυσικά δεν είναι στο ύψο των προσδοκιών μας. Για να εξασφαλίσουμε όμως ότι κανένας δεν θα μείνει ξεχασμένος με βάση την ατζέντα του 2030 και τις ε, δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη, οι FTA θα πρέπει να δημιουργούνται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συμμόρφωση. Όπου τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται αποτελεσματικά και όπου δίδεται υποστήριξη στις τρίτες χώρες επαρκώς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να γίνεται αποτελεσματικά εφαρμογή. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα κεφάλαιο για το φύλλο και την ε, ισότητα των φύλλων σε μια FTA, τότε θα πρέπει διάφοροι εμπλεκόμενοι από τις οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν. Ε, και στο διάλογο, ας πούμε, για τη συμφωνία με τη Χιλή, να καλέσουμε και τους σχετικούς φορείς για να δούμε τι θέλει η Χιλή και αν θέλει τα ίδια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από το Επίσης ε, υπάρχουν οι μεγαλοπεριφέρειες. Εμείς θέτουμε τα πρότυπα πέρα από τις ε, κοινωνικές αξίες ε, και σε άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στο μηχανισμό επίλυση διαφορών επενδύσεων κρατών. Καθώς θα προχωρούμε και θα γίνει υπουργική το Δεκέμβριο του ΠΟΕ, ελπίζω να υπάρξει αλλαγή στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εταίρους, ούτως ώστε η εμπορική πολιτική που θα προωθηθεί να είναι για το κοινό καλό και να δημιουργήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση ακαδημαϊκού χαρακτήρα σχετικά με την εμπορική πολιτική. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Και θα ξεκινήσω με τους συντονιστές. Ο καθένας έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του. Η συνάδελφος Δόκια Σάιφ θα πάρει το λόγο στη θέση μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ σε όλους εσάς για τις παρουσιάσεις σας. Ακούσαμε προσεκτικά όσα είπατε και αργότερα θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια συμπεράσματα σχετικά με αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση της εμπορικής στρατηγικής. Προς το παρόν θα ήθελα να εστιάσω, κύριε Επίτροπε, στις διμερείς συμφωνίες και συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Πρόκειται για ένα θέμα που επανέρχεται τακτικά, μας απευθύνουν συχνά ερωτήσεις σχετικά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ανησυχούν σχετικά με τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν σκοπεύει να αναπτύξει συγκεκριμένη μέσα που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υποφεληθούν περισσότερο από τις συμφωνίες και προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες έχετε ε, αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα επειδή κάποιες πτυχές των συμφωνιών δεν ε, εφαρμόζονται. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω τον λόγο, η κυρία Μόσκα. Και εγώ θεωρώ ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να θεωρήσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Όμως ε, το θέμα είναι να είναι συνεπείς οι πολιτικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι καλό λοιπόν που για πρώτη φορά που μπήκαν στις συμφωνίες και η περιβαλλοντική πολιτική και η διάσταση της ισότητας των φύλων, γιατί η εμπορική πολιτική μπορεί να είναι ένας επιταχυντής και ένας καταλήτης άλλων πολιτικών, που θεωρούμε σημαντικές για να ενισχύσουμε ένα σύστημα αξιών και ευημερίας σε όλο τον κόσμο. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα μόνο θέμα από όλα από όλα όσα ακούσαμε. Το θέμα της παρακολούθησης. Έτσι. Εφαρμογή δηλαδή και παρακολούθηση. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες τίθενται σε ισχύ. Τι γίνεται. Είναι σημαντικό να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση. Γιατί δίδονται κάποιες υποσχέσεις ε, στα πλαίσια των συμφωνιών. Να δούμε λοιπόν Πού φτάσαμε. Επομένω, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, ούτω ώστε κάποιε χώρε που έχουν εμπορικέ συμφωνίε με εμά να μην προωθούν παρόλα αυτά πολιτικέ οι οποίε ε, μειώνουν τα πιθανά ωφέλη. Παραδείγματο χάρη, είδαμε τα παραδείγματα με τον Καναδά τέτοιου τύπου. Με το Βιετνάμ επίση. Δεν έχει επικυρωθεί βέβαια ακόμα η συμφωνία. Υπάρχουν όμω τάσει που μπορεί να μειώσουν τα ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τι εμπορικέ συμφωνίε. Ευχαριστώ πολύ σε όλους τους ομιλητές. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις προσδοκίες σας και τις ε, ελπίδες σας σχετικά με την ε, εμπορική πολιτική και τους σχετικούς κανόνες. Θα ήθελα όμως να ακούσω κάτι παραπάνω από το κύριο Ρότιν και την κυρία Γκαμάς και ε, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου κατά κάποιο τρόπο. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. η βελτίωση, πρόκειται για αντιπαράθεση ανάμεσα στους καλούς και τους κακούς κανόνες εμπορικής πολιτικής ή βρισκόμαστε σε μια θέση όπου έχουμε επιλογή ανάμεσα στους κανόνες και στην απουσία κανόνων. Γιατί βλέπω κάποιους οικονομικούς φορείς να αναπτύσσονται οικονομικά, να αναπτύσσονται και οι φιλοδεξίες τους. Θα θέλαμε πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εντείνει τις απαιτήσει της ε, απέναντι στους εμπορικούς εταίρους. Η δεύτερη ερώτηση είναι εξής σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική. Πολλοί ανησυχούν ιδιαίτερα ότι θα αλλάξουμε την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσα από τις ε, συμφωνίες. Για παράδειγμα, στο τομέα της προστασίας των προσωπικών ε, δεδομένων. Και πάντα τους καθησυχάζουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν ε, αποτελούν μέσο για την τροποποίηση της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτές τις ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνήθως στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων υπάρχουν δύο πιο ακραίες αν θέλετε Θέσει ε, Η μία δηλαδή που μας λέει να εστιάζουμε περισσότερο στο εμπόριο, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα εμπόδια στην αγορά, τους δασμού, ε, τα μη δασμολογικού χαρακτήρα εργαλεία, τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, δηλαδή τεχνικά ζητήματα, ενώ η άλλη άποψη είναι εκείνη η οποία ε, θέλει τη συμπερίληψη όλων και περισσότερων μη εμπορικών στοιχείων, δηλαδή ε, προστασία του περιβάλλοντος, εργασιακά δικαιώματα και άλλα ε, ζητήματα. Άρα λοιπόν ναι, το ποια από αυτές τις δύο στάσεις υιοθετούμε εξαρτάται βέβαια και από την πολιτική μας στάση τελικά, από την πολιτική μας θέση και κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε σε μια χρυσή τομή, σε ένα συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως οι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου μπορούν να είναι και καθώ αναφέρθηκε σε δύο συγκεκριμένε περιπτώσει επίτροπου, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ω προ το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την Ιαπωνία. Καθώ ε, θεωρώ πω είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Και δεύτερο, ε, θεωρείτε πω ε, είναι δυνατόν να ε, ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με ε, τι ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Κύριο Σόλτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, Πρόεδρε, όλους τους ε, ομιλητές ε, όσα μας είπαν. Και ο Σαμπλουτσίνη μας είπε ότι το εμπόριο θα πρέπει να διασφαλίζει καλύτερης ποιότητας, φθηνότερα, πιο ε, προσβάσιμα προϊόντα. Αλλά ποιος είναι εκείνος που θα αποφασίζει ποια είναι τα φθηνότερα, ποια είναι τα καλύτερα, ποια είναι τα πιο προσβάσιμα προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Εσείς μας είπατε ότι θα πρέπει να δούμε το εμπόριο ως εργαλείο. Κατά συνέπεια θα πρέπει να συγκρίνουμε το ποιες είναι οι συνθήκες ε, αυτού του εμπορίου και τι συνεπάγεται αυτό σε ό,τι αφορά τους ε, πολίτες μας, τις κοινωνίες μας, τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε, όταν κάνουμε λόγο για το εμπόριο για όλους, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτή την πτυχή. Δηλαδή, ποιο υποφελείται από αυτό, από την αγορά δηλαδή ενός ε, προϊόντος και αυτό το προϊόν που παράγεται και με ποιο κόστος. Και μου άρεσε πολύ η προσέγγιση που ακολούθησε η Επίτροπος όταν αναφέρθηκε ε, στην έννοια ε, του δίκαιου εμπορίου, του fair trade, μέσα σε αυτήν τη στατική του εμπορίου για όλους. Δηλαδή θα πρέπει να αποτελέσει, αν θέλετε, ε, το, τη, μονάδα μέτρησης ή το, το, υπόδειγμα με βάση το οποίο θα κρίνουμε ότι ναι, το εμπόριο θα πρέπει να είναι φθηνότερο για όλους. Δηλαδή θα πρέπει να είναι φθηνότερο και για τον καταναλωτή, αλλά θα είναι και το φθηνότερο και το καλύτερο απλώ ποιότητα και για το, το, περιβάλλον. Άρα σε ό,τι αφορά την παγκόσμια αλυσίδα αξία και τη στρατηγική ε, εμπόδιο για όλου, αυτά τα δύο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ του. Κύριε Ροντρίγκε Πινίδο, τώρα το λόγο. Perdón, pero eh, va, va con retraso la traducción. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές του πάνελ για τις παρεμβάσεις τους ειδικά την Επίτροπο για την προσπάθειά της για να προωθηθεί σε πολυμερές επίπεδο η οδηγία για τα όργανα βασανισμού, για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων κτλ. Αλλά πέραν αυτών θέλουμε και κάτι άλλο. Αυτές οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου θα πρέπει να ενέχουν και μία δέσμευση ότι όλα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και για αντιθανατική ποινή δεν μπορούν να ε, μπουν στο εμπόριο, να τα εμπορευτούμε ε, με τους εταίρους μας. Θα πρέπει να απαγορευτεί αυτό. Τώρα, για τις ε, δασμολογικές ποσοστώσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Γκαμάζ, ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε τρίτες χώρες ε, που είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένε από εμά έχουν πάρα πολλέ δυσκολίε να σεβαστούν την τεχνική νομοθεσία που απαιτούμε εμεί και που προασπιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν λέω να μειώσουμε τα πρότυπά μα, αλλά να συντονίσουμε την συνεργασία μα ούτω ώστε να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει των τρίτων χωρών που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε να υποφεληθούν και αυτέ από το εμπόριο. Τέλο, η εφαρμογή. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να απαιτήσουμε ότι αυτό που γράφουμε το εφαρμόζουμε κιόλα. Και οι κανόνες για τα εργασιακά δικαιώματα να μπαίνουν ε, και στις ε, εμπορικές συμφωνίες. Λέει κυρία Μίνερ. Έχω διάφορες ερωτήσεις, Πρόεδρε. Θα βγάλω και λίγες ε, από τον κατάλογό μου, αλλά η ΣΕΤΑ δεν νομίζω ότι είναι πρότυπο για τις συμφωνίες ε, ελευθερου εμπορίου, γιατί είναι, υπολείπεται από τις FTA. Δεν θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να αναθεωρήσει τα πράγματα. Υπάρχει μια μελέτη που εκδόθηκε χθες από τους φίλους της γης, τη ΣΥΛ και το δίκτυο των Βρυξελών για τα περιβαλλοντικά με σκληρές κριτικές για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, για, το... για πολυμερείς συζητήσεις και τον τρόπο που διεξάγονται. Υπάρχουν θέλω να ακούσω ε, αντιδράσεις της Κομισιόν για τη μελέτη αυτή και τις επιπτώσεις ε, στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών ε, επενδύσεων, μεταξύ επενδυτών και κρατών. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Όλοι συμφωνούμε ότι η εμπορική πολιτική είναι ένα εργαλείο αλλά γιατί, για το περιβάλλον, για τα εργασιακά, για τους κανόνες, και ελπίζω και για τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες, γιατί θα πρέπει να εξυπηρετεί και τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η εφαρμογή υπό όμως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, είναι μια προϋπόθεση. Ε, μ' αρέσει η έκθεση της Επιτροπής για την Εφαρμογή, τη χαιρετίζω, είναι πολύ σημαντική. Ποιος είναι ο ρόλος όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε όλα αυτά, γιατί στη φάση της, του, της εφαρμογής καλό θα ήταν να παίξουμε πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Ε, Ούτω ή άλλω η συνθήκη τη Λισαβόνα μα έδωσε μεγαλύτερο ρόλο στην εμπορική πολιτική και στην εμπορική δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Και έχουμε διάφορα εργαλεία, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε ε, ομάδε παρακολούθηση, έχουμε τη συμμετοχή μέσω εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να οικοδομήσει ένα διαρθωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με συμβουλευτικές ομάδες, με διπλωματικούς κύκλους από τρίτες χώρες. Το ερώτημα είναι, εσείς πώς το βλέπετε. Μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας. Καταρχάς μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν ναι, μπορούμε να συμμετάσχουμε περισσότερο ή καλύτερα ως κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτ έθεσε ένα ερώτημα. Ποιο αποφασίζει τι είναι πιο φθηνό και τι είναι καλύτερο. Να σου απαντήσω, κύριε Σόλτ. Όλοι μα ως άτομα και ω καταναλωτέ. Αυτό είναι το υπέροχο με την οικονομία τη αγορά. Είναι εθελοντική, δημοκρατική, αποκεντρωμένη προσέγγιση. Το δικό μου ερώτημα αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ζητείτε ε, ένα κεφάλαιο πιο πλούσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που να εφαρμόζεται. Εγώ δεν λέω ότι το κεφάλαιο που έχουμε τώρα δεν εφαρμόζεται, αλλά πέραν αυτού θέλω να σας πω το εξής, να σας ρωτήσω κάτι που είναι το εξής. Από ποιο θα μάθουμε εμείς. Πριν μου πείτε από τους Αμερικάνους, να σας πω, δώστε μου ένα παράδειγμα ε, για το πότε η Αμερική χρησιμοποίησε αυτά τα υπέροχα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και πριν μου απαντήσετε απέναντι στη Γουατεμάλα, να μου πείτε αν μπόρεσε να τα χρησιμοποιήσει νόμιμα αυτά τα κεφάλαια εναντίον της Γουατεμάλας ή τα χρησιμοποιει σε παράνομα. And ευχαριστώ. Αντίθετα με αυτά που είπαν καποιοι από τα μέλη του πάνελ, θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επιτυχής. Νομίζω ότι έχουμε ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο ε, στο εμπόριο με τις ε, υπηρεσίες για τα γεωργικά προϊόντα και γενικά για τα αγαθά. Έχουμε την ε, ρήτρα για, τα, τη δημοκρατία, την βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Όλα αυτά είναι θετικά. Δύο ερωτήσεις. Ένα προς την Επίτροπο. Ξέρετε πολύ καλά τις απόψεις μου εμείς ε, ε, έχουμε καθυστερήσει, ε, με τον Καναδά καθυστερήσαμε 7 χρόνια, σήμερα το πρωί είχαμε το Μερκοσούρ. Πώς θα βελτιώσουμε το χρόνο αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ερώτηση για τον προστατευτισμό. Η κυρία Ντεπινιέρο σήμερα το πρωί μίλησε για τα προστατευτικά μέτρα εναντίον ενό προϊόντο ενό κράτου μέλου που υιοθέτησαν τρίτε χώρε. Πώ θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε, να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε με τι Ηνωμένε Πολιτείε. όταν εμεί οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου ΕΠ και του παγκόσμιου εμπορίου. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές μας. Ε, ευχαριστήσω τον Επίτροπο Άμστροπ. Είμαστε ευχαριστημένοι με τα επιτεύγματά μας σε ό,τι αφορά δηλαδή τις σύγχρονες συμφωνίες που έχουμε επιτύχει σε ό,τι αφορά την Απονία, τον Καναδά και άλλους. σε ό,τι αφορά τους κανόνες στους οποίους αναφερθήκατε είπατε ότι επιβάλλουμε την τήρηση αυτών των κανόνων στους εταίρους μας και ακριβώς μέσω της τήρησης των κανόνων του ΠΟΕΟ. Ωστόσο, δεν αναφερθήκατε στην περίπτωση της Κίνας, κύριε Επίτροπε. Και τη στρατηγική της Κίνας, One Road, One Belt, ένας δρόμος, μία ζώνη, που αποτελεί βέβαια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Η Κίνα δηλαδή ε, ακολουθεί τελείως ε, δικούς της κανόνες, ε, προβαίνει δηλαδή σε στην εξαγορά ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων ε, και στις υποδομές αλλά και ε, στον, σε καινοτόμου τομεί ε, και σε αυτών των προφοριών τεχνολογίας. Και αν λάβουμε υπόψη μας πως οι επενδύσεις της Κίνας σε ένα μόνο μέλος στη Γερμανία δηλαδή από το 2015 προς το 2016 αυξήθηκε πάρα πολύ και έφτασε στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ καταδεικνύει το πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την Κίνα. Οπότε, ποιο θα είναι ο αντίκτυπο αυτή τη εμπορική πολιτική τη Κίνα στη δική μα. Γιατί βέβαια η επενδυτική πολιτική αποτελεί αναπόσταστο τμήμα τη εμπορική μα πολιτική. Σήμερα το πρωί εμεί συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή ε, την διαδικασία ελέγχου των εξαίρων επενδύσεων. Μήπω ε, μια τέτοια διαδικασία έρχεται πολύ καθυστερημένα και δεν επαρκεί. Κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου στη σελίδα 32 αναφέρει ότι θα συνταχθεί ο δικός χάρτης. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Θα καλύψει ο δικός χάρτης την βιώσιμη ανάπτυξη και δεύτερον όπως είπε και ο κύριος Βίνκλερ, θα σταλεί στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, επικύρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρη στη διαφάνεια. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω σε έναν συνάδελφο που είχε τη τάση να περιορίζει τη συζήτηση για το εμπόριο την ιδεολογική τοποθέτηση κάποιων ε, προοδευτικών και κάποιων συντηρητικών. Είναι σαν καρικατούρα. Δεν συμφωνώ καθόλου με μια τέτοια θέση, εκτός αν ε, θεωρούμε ότι οι προοδευτικοί ε, ακολουθούν μια συνεκτικότητα, οι συντηρητικοί όμως όχι. Διαφορετικά, αν, μιας και βρισκόμαστε στα πλαίσια συμφωνιών, εμπορικών συμφωνιών, όλο ένα και πιο με όλο ένα μεγαλύτερο εύρος. Οπότε είτε πρόκειται για τη διανοητική ιδιοκτησία είτε για το δικαίωμα ρύθμισης είναι σημαντικό να προβλέπονται τα αντίστοιχα μέσα. Όταν μιλάμε για δασμού είναι απλό, όταν μιλάμε όμως για εναρμόνιση των κανόνων τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Είναι απαραίτητη μια ισορροπία των δυνάμεων. Και εγώ θέτω το εξή ερώτημα. Γιατί να προστατεύσουμε επενδύσεις και γιατί να μην προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί σε τέτοιες συμφωνίες δεν προστατεύουμε το δικαίωμα ε, της πρόσβασης στο περιβάλλοντος. Δεν είμαστε κατά της προστασίας των επενδύσεων, αλλά σήμερα έχουμε πολύ ανισόρροπες συμφωνίες. Αν επανέλθουμε σε μια ισορροπημένη προσέγγιση στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών, θα είναι όλα πολύ πιο απλά για όλους και δεν θα συμμετέχουμε σε μια ιδεολογική συζήτηση όπως προσπαθούν κάποιοι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις από το Twitter. Ε, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την υγεία των ζώων. Και δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ε, δυσκολίες ε, στους κόλπους του ΠΟΗ και τις ε, διμερείς συμφωνίες. Από την άποψή μου, το 70% αφορά την παγκόσμια λυσίδα αξίας. Δεν θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτήν από το να προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις συμφωνίες με κάποια χώρα. Και τώρα δίνω το λόγο Στην Επίτροπο έχετε τέσσερα λεπτά. Be very brief because I wanted also to respond to... Ναι, ε, πολύ σύντομα. Ήθελα να απαντήσω στις κάποιους από τους άλλους ομιλητές, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ γρήγορα. Ε, ε, προφανώς το εμπόριο αφορά τους ανθρώπους του και, και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, ε, και η μεγαλύτερη ανισότητα, αν θέλετε, που ισχύει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν μια θέση εργασίας και τους ανέργους. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ανισότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει ακριβώς μέσω του εμπορίου να το επιτύχουμε. Ε, ε, δηλαδή ε, μέσω των εμπορικών συμφωνιών δημιουργούμε θέσει εργασία με καλύτερου μισθού και καλύτερε εξειδικεύσει. Και βέβαια αυτέ τι θέσει εργασία υφίστανται στι επιχειρήσει. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Οι επιχειρήσεις δηλαδή δίνουν εργασία στους πολίτες. Από εκεί και μετά μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει δηλαδή να δραστηριοποιηθούν πολύ περισσότερο στο πλαίσιο των οργανώσεων μικρομεσών επιχειρήσεών τους. Εμείς δηλαδή παρέχουμε πολύ καθοδήγηση, πληροφορίες, καλά παραδείγματα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα σχετικά κεφάλαια. στι ε, συμφωνίε ελεύθερο εμπόριο. Και έχουμε ε, εξετάσει το ενδεχόμενο του να δημιουργήσουμε ειδικέ, αποκλειστικά δηλαδή για μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, ιστοσελίδε. Και αυτά τα ζητήματα τα συζητάμε και με διαφορετικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια ε, και με τι ε, χώρε εταίρου μα Τώρα σε ό,τι αφορά του κανόνε προέλευσης, ναι, είναι υπερβολικά περίπλοκοι και προσπαθούμε να επιτύχουμε μια απλούστευση, ειδικότερα στο πλαίσιο τη Μεσογειακή Συμφωνία, τη Euromed δηλαδή, αλλά εδώ θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, σίγουρα. Παρότι βέβαια παραμένει εξαιρετικά περίπλοκος, περίπλοκο αυτό το ζήτημα, θα γίνει κάτι. Χωρί να μπορώ να σα υποσχεθώ ότι κάτι θα γίνει πολύ σύντομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα με την Ιαπωνία, νομίζω πω θα φτάσουμε εδώ πολύ ε, γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα, το Δεκέμβριο δηλαδή. Υπάρχουν κάποια τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα και το μόνο πολιτικό ζήτημα ε, που παραμένει εκρεμέ είναι το πώ αντιμετωπίζουμε την προστασία των επενδύσεων. Δηλαδή το ε, δικό μα νέο σύστημα δημιουργεί μια διαφοροποίηση καθώς οι Ιάπωνες θεωρούν ε, πως το παλαιότερο σύστημα ήταν πολύ καλό αλλά χωρίς να υπάρχει ε, τόσο μεγάλο ύψος ε, να επενδύσεων μεταξύ των δύο μπλοκ δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την, τις ΗΠΑ και το αν θα μπορούσαν να επανεκκινηθούν ή όχι είναι ορατό στο, στο μέλλον αλλά δεν γνώριζουμε πότε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων, capacity building στι αναπτυσσόμενε χώρε, ναι, το κάνουμε έτσι, ώστε να μπορέσουν και εκείνε να αξιοποιήσουν περισσότερο ε, ε, τις, ε, διεθνείς αγορές, ειδικότερα μέσω τη ανάπτυξη των υποδομών του. Ε, και ε, ένα μεγάλο τμήμα τη αναπτυξιακή βοήθεια που κατευθύνεται προ αυτέ τι χώρε, ακριβώ αφορά την δημιουργία αυτών των υποδομών. καθώ το εμπόριο και η ανάπτυξη κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Τώρα σε ό,τι αφορά το Friends of the World και τη, σχετική έκθεση ναι, ε, ε, δεν νομίζω πως ε, είναι πολύ, μας εκπλήσουν πολύ αυτά τα αποτελέσματα. Δεν έχω ενθουσιαστεί ιδιαίτερα. Δηλαδή για 15 εβδομάδε υπήρχαν τα σχετικά έγγραφα διαθέσιμα για την υποβολή σχολείων. Και ανταλλαγή απόψεων, οπότε οι Friends of the Earth είχαν σε, όλες αυτές, σε όλη αυτή την περίοδο τη δυνατότητα να αποστείλουν τα σχόλιά τους. Υπήρξαν δημόσιες ε, ε, συζητήσεις, η έκθεση σε ό,τι αφορά τη δημόσια διαβούλευση είναι και εκείνη δημοσίως ε, Διαθέσιμο οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώ μα λένε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ε, ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να είναι επίσημο, δεν νομίζω πω θα ήταν χρήσιμο όταν είναι επίσημο, αλλά ανεπίσημο ναι. Γιατί έχετε τι δικέ σα διακοινοβουλευτικέ ε, επιτροπέ, ακούτε μία σειρά από πληροφορίε, ακούτε ω προ το ποια στοιχεία είναι εκείνα που λειτουργούν καλά και ποια λιγότερο καλά. Και τέτοιου είδου πληροφορίε θα μπορούσαν να ήταν εξαιρετικά χρήσιμε για την Επιτροπή, αν μα τι διαβιβάσετε στο επίπεδο τη εφαρμογή. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε δηλαδή κάποιε ειδικέ επιτροπέ σε αυτά τα ζητήματα. Προφανώ εξαρτάται από εσά. Αλλά σε ό,τι αφορά την επίσημη εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών, δεν νομίζω πω θα έπρεπε να αναλάβει ένα επίσημο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, ε, κύριε Σαλαφράκα, ναι, πράγματι ε, είναι χρονοβόρα η εφαρμογή τέτοιων ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να. Ε, πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε καχύνουμε τέτοιου είδου διαδικασίε. Για παράδειγμα, αν η κύρωση στο μέλλον χρειαζόταν να γίνει όχι από τα εκάστοτε κράτη-μέλη, αλλά από το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω θα μπορούσαμε να είχαμε μια ταχύτερη διαδικασία. Και επίση γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα των ελιών που έχει προκύψει και συνεργαζόμαστε στενά με την Ισπανική κυβέρνηση αλλά και την Περιφερειακή κυβέρνηση τη Ανταλουσία, προκειμένου να μην ε, προβεί στα όσα έχει απειλήσει να κάνει η Αμερικανική πλευρά. Πάντω, ήδη το πρώτο βήμα που έχει λάβει δεν είναι, είναι δυσανάλογο, οπότε θα ε, συνεργαζόμαστε όσο ε, περισσότερο μπορούμε με την Ισπανία. Τώρα, η Κίνα αποτελεί μια ε, πρόκληση, αποτελεί ένα δυνητικό εταίρο, αλλά δύσκολο ε, ε, εταίρο και βέβαια οι επενδύσει τη Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προβληματικές από τη φύση τους. Απλώς σχετίζονται με το κατά πόσο συνδέονται και με κάποιες πολιτικές συνθήκες. Γι' αυτό, γι αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, αυτή την πλατφόρμα σε ό,τι αφορά τον, την παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων προκειμένου να υπάρχει μια καθοδήγηση, γιατί βέβαια πρόκειται για ένα τοξικό ζήτημα στο Συμβούλιο, γιατί βέβαια εσεί μα είπατε πω ένα τέτοιο εργαλείο του ελέγχου των ε, ε, επενδύσεων είναι πολύ αδύναμο, ενώ τα μισά κράτη στο Συμβούλιο θεωρούν ότι είναι υπερβολικά ισχυρό ήδη. Α δούμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και στο εξή επίπεδο τη εφαρμογή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χάρτη πορεία στο roadmap, ε, θεωρώ ναι, πω θα δημοσιευτεί. Θα το ελέγξω, αλλά ναι, νομίζω πω θα είναι δημόσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευμερία των ζώων. Ναι, αναφερόμαστε εδώ στα διεθνή πρότυπα και στις ε, διεθνείς συνθήκες ε, και ε, προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε κάτι παραπάνω εδώ στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Μεξικό, αλλά και με άλλες χώρες. Βέβαια το βασικό ζητούμενο είναι εδώ να αρχίσουν να συνεργάζονται μαζί μας οι διάφοροι εταίροι στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων που ισχύουν. Και ακούμε πολλά σε σχέση με την ευημερία των ζώων ε, από διάφορες οργανώσεις οι οποίες ε, μας ε, έδωσαν κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, άλλες βέβαια λιγότερο. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση. συγγνώμη που αχρηγόρησα, αλλά τα περισσότερα ερωτήματα σχεδόν στέθηκαν σε μένα. Ευχαριστώ. You, mean the body? No, Ρωτάτε. Συζήτηση εκτός μικροφώνου there is not really a in, in the... Υπάρχει μπλοκάρισμα στον ΠΟΕ, αλλά είναι αργή διαδικασία. Γι' αυτό και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος ε, μπερδεύεται με αυτές τις ε, περιφερειακές ή διμερείς συμφωνίες. Ατυχές είναι που μπερδευόμαστε έτσι, αλλά είναι αναπόφευκτο. Γιατί δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα στα πλαίσια του ΠΟΕ με 164 μέλη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει γιατικό ρόλο στη Γενέβη, ούτω ώστε να έχουμε ένα, μια διεθνή πολυμερή συμφωνία και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλες μας συμφωνίες ε, συμμορφούνται με τους κανόνες του ΠΟΕ, αλλά το να περιμένουμε όλους αυτούς τους κανόνες για την απελευθέρωση της ε, αγοράς να περάσουν μέσω του ΠΟΕ, τότε δεν θα είχαμε καθόλου εμπόριο. Ο κύριος Ρέντι. Ευχαριστώ. Είμαι Γερμανός ε, συνδικαλιστής, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, και άρα είμαι πολύ υπέρ του ελευθέρου εμπορίου. Δεν είναι το θέμα αν είναι κανείς κατά υπέρ του ελευθέρου εμπορίου. Το θέμα είναι αν θέλουμε να έχουμε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που είναι υποφελείς για τους ανθρώπους ή όχι. Και εγώ εκπροσωπώ ε, ανθρώπους και κυρίως εργαζόμενους. Άρα θέλουμε να έχουμε ε, ε, τέτοιες συμφωνίες που ενισχύουν και όχι υποσκάπτουν την ποιότητα της εργασίας των θέσεων απασχόλησης και την αξιοπρεπή απασχόληση. Αυτό είναι η πρόκληση. Ακούσαμε τη συζητήση ότι πολλές συμφωνίες είναι πραγματικά αμυγός εμπορικές συμφωνίες. Τώρα όμως προωθούν οι μοντέρνες συμφωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες που είναι δύσκολες. Οι υπηρεσίες ε, είναι εδρασμένες στο εθνικό πλαίσιο και αυτό έχει επιπτώσεις. Και εδώ μιλάμε για τις παγκόσμιες αλυσίδες ε, παροχής, ας πούμε, που, είναι, που παράγουν προϊόντα ε, τα οποία εξάγονται κτλ. Αλλά και στις ε, υπηρεσίες γίνεται το ίδιο με τις παγκόσμιες αλυσίδες. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αδιαφάνεια και το, το, το καθεστώς είναι άμορφο ακόμα. Υπάρχουν πολλές εταιρείε και κυβερνήσεις που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ε, το ότι υπάρχει εκεί, όχι για δίκαιο εμπόριο, αλλά για άδικο εμπόριο. Και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μαζί με τα θεσμικά όργανα στην ε, Ευρώπη υπάρχει δίκαιο εμπόριο που υποστηρίζει την ευημερία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Επίσης, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε και την ευημερία των εργαζομένων στις τρίτες χώρες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη ως ο παγκόσμιος ε, εμπορικός παράγοντας στον κόσμο, ε, αν δεν κάνει αυτή αυτά που πρέπει να κάνει, δεν θα το κάνει κανένας άλλος και σίγουρα δεν θα το κάνει η Κίνα. Άρα έχουμε ευθύνε να προχωρήσουμε. Και πρέπει να πούμε ότι έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, το αν θα πετύχουμε το ιδανικό μοντέλο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το βασικό είναι να πούμε αυτή είναι η στόχη μας. Ε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο optimum. Α προσπαθούμε να συνεργαστούμε ω ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με του κοινωνικού εταίρου, ούτω ώστε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Μερικές φορές, ε, όταν μιλάμε για το εμπόριο, παίζουμε πολύ με ιδεολογήματα. Μιλάμε πολύ με ιδεολογήματα. Το εμπόριο είναι ένα εργαλείο μοναδικό όπου οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα ε, το χρησιμοποιούν Αυτό συνδέεται με πολλά από τα ερωτήματα που άκουσα. Το πρώτο αφορά τα πρότυπα. Η Ευρώπη είναι πρωταθλήτρια στο εμπόριο στην, ε, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο, όχι μόνο στο εμπόριο. Έχουμε ένα μοντέλο οικονομίας που είναι μοναδικό. Και αυτό είναι τμήμα της ταυτότητάς μας. Και αυτό είναι αυτό που εξάγουμε στο εξωτερικό. Δεν έχει νόημα οι επιχειρήσεις ε, να παίζουν ε, με ένα πρόσωπο στην Ευρώπη και με ένα διαβολικό πρόσωπο στο εξωτερικό. Και δεν το κάνουν οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Δεν το κάνουν. Γιατί οι κανόνε και τα διάφορα εργαλεία που έχουμε ε, φτιάξει εδώ και δεκαετίες, για να πω αιώνε στην Ευρώπη, μα εμποδίζουν να λειτουργήσουμε έτσι. Ακριβώ αυτό είναι σημαντικό όταν κάνουμε εμπόριο στο εξωτερικό. Δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση κούρσα προ τα κάτω. Δεν αλλάζουμε τα πρότυπα. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει το θέμα του να προωθήσουμε πράγματα που, δεν έχουν, που είναι περιφρονητέα στις δικές μας κοινωνίες. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν κακοί παντού. Ακόμα και στο δρόμο, ας πούμε, ε, υπάρχουν οδηγοί που παρά τα όρια τρέχουν σαν τρελοί. Και δεν σε τον κόκ. Αλλά Εμείς παίζουμε τους κανόνες. Είμαστε πρωταθλητές και στην πολυμέρεια και στην, στο σεβασμό των προτύπων για την ασφάλεια και την κοινωνική προστασία. Ένα δεύτερο που θέλω να πω. Αφορά την εφαρμογή. Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο στο θέμα της εφαρμογής, το οποίο είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή η Επίτροπος Μάλστρομ ε, υπογράφει τη συμφωνία. Τι γίνεται αμέσως μετά. Φυσικά υπάρχει επικύρωση στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι πώς ε, εμπλέκονται οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες στην προώθηση των αξιών, στο να υπάρξουν ωφέλη, στο να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες. Εκεί μπορούν να κάνουν πολλά οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες. Στην έκθεση εφαρμογή νομίζω ότι δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τι μικρομεσαίέ επιχειρήσει. Όλοι λέμε ότι είναι τόσο σημαντικέ, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, γιατί να μην αντιμετωπίζουμε τις, τα θέματα αυτά από τη σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φερρυπίν, το θέμα τη εφαρμογή, αλλά και το θέμα του δικού χάρτη από τη σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλο, Ποιο θα υποφεληθεί, Ποιο αποφασίζει τι είναι καλό, τι είναι φθηνό, τι είναι διαθέσιμο. Στον επιχειρηματικό κόσμο υπάρχει ένας δικαστής που δεν έχει ίκτο. Είναι η αγορά. Και ποια, ποιος είναι η αγορά? Είναι οι καταναλωτές. Αυτοί μας κρίνουν κάθε μέρα. Λειτουργούμε με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και ο τελικός κριτής αυτού είναι ο καταναλωτής που θα αποφασίσει αν θα αγοράσει ή δεν θα αγοράσει τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Um, Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε κατά της, ε, του ανοιχτού χαρακτήρα των αγορών. Εμείς ε, θέλουμε από τις αγορές, ε, αν θέλουμε να τηρούν οι αγορές κάποιες κοινωνικές δεσμεύσεις, πρέπει να, το, να τις περιστηρίξουμε. Και αυτό αφορά όλες τις διαπραγματεύσεις που, ε, για εμπο, συμφωνίες εμπορικο, ε, ελεύθερου εμπορίου. Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ε, αξιολογήσεων επιπτώσεων κατά διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μετά. Και εκεί που χρειάζεται περισσότερη δουλειά είναι το πώς καθορίζουμε αν μια κατάσταση έχει βελτιωθεί ή όχι ε, από τη στιγμή που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μια συμφωνία και κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση, κοινωνικοί εταίροι, διάφοροι οργανισμοί. Πώς ε, κρίνουμε αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αν τηρούνται οι αξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στόχος μας δεν ήταν να ε, λύσουμε όλα τα προβλήματα. Έχουμε ακούσει ε, πολλά. Ευχαριστώ πολύ σε όλους τους ομιλητές. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο πάνελ και ε, καλώ τους ομιλητές του επόμενου πάνελ να έρθουν να καθίσουν δίπλα μου. Okay, so now we Πολύ ωραία. Ξεκινάμε τη συζήτηση στα πλαίσια του δεύτερου πάνελ με εστίαση στη σχέση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και το εμπόριο. Τίτλος του πάνελ ε, «Το εμπόριο για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης». Έχουμε τέσσερις εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα. Η κυρία Έλεν Βόλφ, ε, ε, αναπληρωτής Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, τον καθηγητή Ιαν Γκόλντιν, καθηγητή εξειδικευμένο στην παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Όξφορντ, την κυρία Κάντζα, υπεύθυνη των περιφερειακών στρατηγικών ε, στο World Economic Forum στη Γενέβη και τον κύριο Κόζουλ Ράιτ, επικεφαλή του Τμήματος Παγκοσμιοποίησης και Στρατηγικών Ανάπτυξης του UNCTAD. Ο κύριος Βόλφ θα αναφερθεί στο ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Χάρηκα πολύ που έμαθα πολλά ακούγοντας τις παρουσιάσεις και τις ερωτήσεις Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω σύντομα στο ρόλο και την αξία του ΠΟΕ και στο τι μπορεί να ακολουθήσει καθώς και στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίηση. Δεν χρειάζεται να ε, γυρίσουμε πολύ πίσω σε ό,τι αφορά την αξία του έργου του ΠΟΕ. Αποδείχτηκε η αξία του ε, μόλις το 2008 ελήφθησαν έκτακτα μέτρα, νομισματικά μέτρα. Δεν ελήφθησαν μέτρα όμως εμπορικού χαρακτήρα, γιατί ακριβώς υπήρχε ο ΠΟΕ και αυτό βοήθησε. Ε, ο ΠΟΕ έχει τέσσερις βασικές δεσμεύσεις, ε, καμία αύξηση των δασμών, καμία επιβολή ποσοστώσεων, απουσία διακρίσεων βάση της χώρας προέλευσης και καμία αρνητική μεταχείριση για τα ξένα προϊόντα και τις ξένες υπηρεσίες. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το σύστημα είναι ικανό να αντιμετωπίσει ε, τις δυσκολίες και τις αναταραχές αντιμετωπίστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η μεγάλη ύφεση. Ο προκάτοχος του ΠΟΕ και ο ΠΟΕ είχαν υπόψη τους ένα σύστημα που θα ήταν ικανό να αντιμετωπίσει οικονομικά ζητήματα και τις επιπτώσεις τους. Σημειώθηκε πρόοδος τα τελευταία χρόνια, η συμφωνία στον Αερόμπι πριν από δύο χρόνια, σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις ε, εξαγωγών, συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, Συμφωνία για τον Πόριο προϊόντα τη τεχνολογία των Πληροφοριών. Δυστυχώ υπάρχουν διαφορές στους κόλπους του ε, ΠΟΕ. Ε, δεν μιλάω σήμερα όμως εξ ονόματο του ΠΟΕ. Έχω όμω τι προσωπικές μου απόψεις, τι οποίες θα μοιραστώ μαζί σα. Το τμήμα παρασχωρήσεων ε, μου υποβάλλει εκθέσεις και σε αυτό το τομέα υπήρχαν ε, σημαντικές επιπτώσεις. Βοσνία, Ρζεγοβίνη, Τιμόρ, Σουδάν, Σομαλία, το Αφγανιστάν και η Λιβερία είναι οι δύο τελευταίες χώρες που προσχώρησαν. Η Λιβερία αντιμετώπισε ε, ε, ε, σύγκρουση και μετά την ε, επιδημία του έμπολα. Όλες αυτές οι χώρες θέλουν πάρα πολύ να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ γιατί πιστεύουν ότι τα χώρια φόρουμ στο οποία εντάχθηκαν για να προσχωρήσουν στο ΠΟΕ θα τους θα ενισχύσει, θα συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. στη Γενέβη επικρατεί μια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Η χώρα που ε, ασκούσε ηγετικό ρόλο και συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικός εταίρος, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω. Μιλάω για τις ε, ΗΠΑ. Δεν φαίνεται να θέλει να ηγηθεί των ε, πολυμερών ε, εγχειρημάτων στους κόλπους του ΠΟΕ και, ε, είναι δύσκολο να υπερβάλλει κανείς ότι δεν θα, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική αναθεώρησης και προσαρμογής σε όλες τις πρωτεύουσες και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, τέσσερις επιλογές. Η μία είναι ένας εθνικός οικονομικός εθνικισμός, για τον οποίο μιλάμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Στόχος είναι τα εμπορικά πλεονεκτήματα ε, για τους εθνικούς παραγωγούς ε, Τέτοιες συμφωνίες ονομάζονται συχνά συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, παρόλο που ε, προβλέπουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά. Η δεύτερη επιλογή είναι η διαπραγμάτευση μιας επιδο... επικοδομητικής συμφωνίας ελεύθερου ε, εμπορίου, που μπορεί να διαμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ε, η ε, εταιρική σχέση του ειρηνικού και η ε, διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Η συμφωνία TTIP δεν είχε στόχο να υπερασπιστεί μόνο το συμφέρον των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών. Η τρίτη επιλογή, η περιφερειακή ολοκλήρωση. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα είναι η ναύτα, η εταιρική σχέση του ειρηνικού, η συμφωνία RCEP. Η ενιαία αγορά βρίσκεται στη μία άκρη του ε, φάσματος και υπάρχουν και άλλες μορφές συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου τέταρτη επιλογή ή ε, σχεδόν παγκόσμιο χαρακτήρα εμπορικές συμφωνίες. Σημασία έχει να ε, εφαρμόζονται οι αρχές όπως η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους ε, και οι σχετικές υποχρεώσεις και η συμφωνία για, περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών δεν τηρείται από όλου. Και η δεύτερη μεγάλη πρόκληση των καιρών μας είναι το τι θα κάνει η ΠΟΕ από εδώ και στο εξής. Τα τελευταία χρόνια, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ μία κατάσταση όπως η σημερινή όπου αποσύρονται οι ΙΠΑ. Πολλά είναι αυτά που μπορούν να κάνουν οι διάφοροι υποψήφοι. Το ε, Brexit ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, και δημιουργεί μεγάλες ενησυχίες ε, το Πεκίνο με τη στρατηγική One Belt One Road, μια ζώνη, ένας δρόμος, το Τόκιο. όπου υπάρχει ανησυχία σχετικά με την εταιρική σχέση ε, του ειρηνικού και η ε, διαπραγματεύση σχετικά με τη Συμφωνία Ναύτα. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το, ε, περίπου το 33% ε, του ε, προϋπολογισμού του ΠΟΕ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει, ε, αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού από τη ΣΥΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία μαζί. Ακόμα και μετά το Brexit. Σημαντικό λοιπόν το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχει ε, μεγάλες δυνατότητες να ηγηθεί του ΠΟΕΠ εδώ και στο εξής βασιζόμενοι μεταξύ άλλων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι το επίπεδο δραστηριοποίηση πρέπει να ενταθεί γιατί οι ΙΠΑ δεν ε, έχουν πια το ρόλο που είχαν στο παρελθόν. Ίσως αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νάψει διμερείς συμφωνίες, ε, μεταξύ άλλων ε, συνεχίζει να διαπραγματεύεται ε, και περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες. 27 συμφωνίες μέτρησα στο, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται όμως αναβάθμιση στους κόλπους του ΠΟΕ, ε, αναβάθμιση προκειμένου να προσαρμοστεί στη ψηφιακή οικονομία και στα διάφορα σχετικά ζητήματα που προκύπτουν πρέπει να προσαρμοστεί στη Συμφωνία για το Εμπόριο Προϊόντων της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και για πολλούς λόγους το ΟΠΟΕ πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Απευθύνω λοιπόν μία έκκληση σήμερα το, και στους, ε, στην Κίνα και στην Ιαπωνία Χρειάζεται μια αναθεώρηση και χρειάζονται ε, επιπλέον προσπάθειες προκειμένου να εξελιχθεί το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόλντιν, καθηγητής Γκόλντιν. Κάτι την απόψή σας. Η στρατηγική εμπόριο για όλους είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιήσει κανείς για να διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση. Καταρχάς, να συγχαρώ την Επίτροπο Μάλστρομ και τους συναδέλφους της για αυτό που κατά την άποψή μου αποτελεί μοντέλο για το τι πρέπει να μοιάζει μια στρατηγική. Και μας πάει πιο πέρα προς ένα πιο υπεύθυνο ε, εμπόριο και επενδυτική πολιτική. Με βάση την πρόσφατη λακωνική αλλά πολύ ενδελεχή έκθεση για το, με τίτλο «Δαμάζοντας την παγκοσμιοποίηση», νομίζω ότι η Κομισιόν θέτει το σωστό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση, σωστό είναι, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες της εμπορική πολιτικής, ε, αλλά θα πρέπει να ε, ειδωθούν αυτές οι ανάγκες σε ένα ευρύ πλαίσιο. Η ΕΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρούν και δεν παίζουν πια ηγετικό ρόλο και δίνεται ο ρόλο τη Κίνα. Την ίδια στιγμή ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο σημαντικό. Επομένω, ο ηγετικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Και όλοι όσοι πιστεύουν, γιατί άκουσα όλου του ομιλητέ και την Κομισιόν να λένε ότι το εμπόριο είναι μια ατμομηχανή όχι μόνο για θέσει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά και για μια καλύτερη ζωή για του τους πολίτες όλου του κόσμου, εφόσον το πιστεύουμε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να το υλοποιήσει αυτό. Αυτό που είναι ανησυχητικό με την αποχώρηση κάποιων χωρών από το εμπόριο, που πηγαίνουν που απομονώνονται και γίνονται πιο προστατευτικές, ε, δεν είναι μόνο το θέμα του τι γίνεται στο εμπόριο. Μέσω του εμπορίου είναι ότι μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να καταλαβαίνουμε τι προτιμήσει μα και να διαπραγματευόμαστε και να φτάνουμε σε κοινά συλλογικά αποτελέσματα. Όταν τα υποσκάπτουμε αυτά, υποσκάπτουμε την ανάγκη μα να δουλεύουμε πάνω σε πολλού άλλου τομεί, Όλο και πιο ε, περίπλοκα παγκόσμια αγαθά. Φέρει πίν κλιματική αλλαγή, μικροβιακή αντίσταση και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να μα απασχολήσουν από κοινού. Άρα το θέμα πάει πέρα από το εμπόριο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό σύστημα που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες παγκοσμίω. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι χώρες του κόσμου και ακόμα και μια μεγάλη περιοχή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το τι κάνουν οι άλλοι και πώς ανταποκρίνονται οι άλλοι και το κατά πόσο για, το, για να μπορέσουμε και εμείς να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον, τον μέλλον μας. Ε, αυτό ισχύει και στην ε, τεχνητή νοημοσύνη, στο γονιδίωμα, στην, ε, στις μηχανές μάθησης κτλ. Έχουμε όλο και πιο περίπλοκα συστήματα. Το 1 τρίτο των θέσεων της απασχο... Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργούνται από το εμπόριο και το μέλλον μας εξαρτάται από το μέλλον των υπολείπων ή αναπτύσσονται οι αναπτυσσόμενες ε, αγορές και έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων αγορών, θεωρούμε ότι το 70% της παγκόσμιας οικονομίας σε 25 χρόνια θα προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές. Ε, και χωρίς αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης ε, στην παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια οικονομία γενικά θα βαλτώσει με τρόπους που θα, που θα κάνουν την χρηματοπιστωτική κρίση να μοιάζει αστεία. Είναι όλα αυτά πολύ θετικά για μας. όσο γινόμαστε πιο πλούσιοι, η ποιότητα της ανάπτυξης θα έχει μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό ισχύει και για την Κίνα, αλλά και για μας. Ε, έχουμε όλο και χαμηλότερους δασμούς. Ε, το βασικό θέμα είναι από εδώ και πέρα οι πολιτικές προτιμήσεις, η ποιότητα, η ποσότητα και πώς θέλουμε αυτές να ενσωματωθούν στα εμπορικά προϊόντα. Ε, οι αξίες μας δηλαδή. Ε, όσο ο κόσμος θα, αποϊλοποιείται, θα γίνεται πιο ψηφιακός, θα πηγαίνουμε σε λογισμικά που θα αποφασίζουν για διάφορα πράγματα όλες αυτές οι επιλογές ε, ε, ενσωματωμένες σε αλγόριθμους θα είναι ένα παράδειγμα για το πόσο γρήγορα αλλάζει το εμπόριο και οι τεχνολογικές αλλαγές θα αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και θα απαιτούν άλλα πράγματα από μας. Επίσης, ε, ένας άλλος τομέας με νέες απαιτήσει είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως την δυνατότητα να δαμάσουμε το γονιδίωμα, ε, πώς αυτό θα επηρεάσει τα έμβρια κτλ. Φυσικά έχουν σημασία όλα αυτά. Τώρα, το αν θα βάλουμε προτιμήσεις για το περιεχόμενο, ας πούμε, του άνθρακα, ε, αυτό θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο. Ε, θα πρέπει επίσης όλα αυτά να, έχουν, να ενσωματώνονται ας πούμε στην εμπορική μας πολιτική. Θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση, περιβάλλον κτλ. θα έχουν σημασία στο εμπόριο για όλους. Ε, και αυτό έχει σημασία όχι μόνο στα φυσικά προϊόντα και στις υπηρεσίες, αλλά και στα ψηφιακά προϊόντα. Ο κόσμος θα αλλάζει όλο και πιο γρήγορα. θα είναι πολύ πιο θα έχει περισσότερες προκλήσεις. Περισσότερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για όλες τις χώρες. Το πώς θα εξασφαλίσουμε διαδικασίες που θα αποκλείουν κανέναν. Ε, οι δυναμικές πόλεις θα αλλάζουν όλο και πιο πολύ και θα είναι πιο ευνοϊκές προς την παγκοσμιοποίηση. Ε, πολιτικές απαντήσεις, πιο ψήφισε για τον Τραμπ, ποιος ψήφισε για τον Brexit, ε, ποιος ψηφίζει την άκρα δεξιά ε, στην Ευρώπη. Ε, αυτοί που ψηφίζουν έτσι δεν είναι αυτοί που υποφελούνται από το εμπόριο, είναι αυτοί που είναι οι ξεχασμένοι, ε, οι εγκαταλελειμμένοι, εγκαταλελειμμένοι γιατί δεν συνδέονται με τις δυναμικές πόλεις. Η, κινητικότητα, ε, το εισόδημα του, του καθενός, ε, όλα αυτά εξαρτώνται από τη σχέση που έχουμε με τις δυναμικές πόλεις. Ε, επίσης, οι νέοι, ας πούμε, από τα... Από κάποιες περιοχές της Αγγλίας, ας πούμε, θα έχουν πολύ λιγότερε δυνατότητε από, ε, από τους γονείς τους να πάνε στη Γαλλία ή σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ε, θα πρέπει οι νέες πολιτικές να δίνουν δυνατότητα στους ανθρώπους να πάνε προς περιοχές όπου υπάρχουν δυναμικές θέσει απασχόλησης. Οι αλλαγές θα είναι όλο και πιο γρήγορες και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το ποιοι είναι οι ξεχασμένοι από αυτές τις αξίες, από αυτόν τον κόσμο αν τους ξεχάσουμε θα κινηθούν αντίον τη παγκοσμιοποίηση, και αυτό το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο. Η ευθύνη μα λοιπόν δεν είναι μόνο απέναντι στο εμπόριο ως ε, στοιχείο μεταρρύθμισης και να εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματικές εμπορικές πολιτικές. Ε, ο ρόλος μας είναι στις πόλεις μας και στους διάφορους τομείς να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια τα, θέματα θα είναι πιο περίπλοκα, ε, οι ανάγκες και δεξιότητες πιο απαιτητικές. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Είναι σημαντικό να κατανοούμε καλύτερα και τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι ε, στην ολοκλήρωση και ενσωμάτωση, αλλά θα πρέπει να του αντιμετωπίσουμε ούτω ώστε τα ωφέλη να αφορούν περισσότερου ανθρώπου πιο γρήγορα και πιο ευρέω. Το ελπίζουμε κι εμεί ότι μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Η Αφρική τώρα ε, αποτελούσε ένα μέρος του κόσμου το οποίο έχει ξεκαστεί για πολύ καιρό. Ενώ ε, κατά τελευταία χρόνια τώρα έχει έλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εδώ του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, η σοσιαλιστική ομάδα οργάνωσε για δεύτερη φορά και αυτή την εβδομάδα τρέχει, δεύτερη λοιπόν Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αφρική. που αφορά ακριβώς και το πώς θα ορίσουμε την πολιτική μα σε σχέση με την Αφρική. Κυρία Κάντζα, λοιπόν, ποια είναι η δική σας ε, άποψη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε ε, και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ καθώς έβλεπα και πέρσι πάλι εδώ στο πλαίσιο της Δημοσίου Ακρόασης και αποτελεί τιμή για μας να έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε μαζί σας την ε, συμμετοχή μας εδώ ε, και την υποστήριξή μας απέναντι στην ε, πολιτική σας ε, trade for all, το εμπόριο για όλους. Επιτρέψτε μου να σας πω το γιατί θεωρούμε σημαντική εμάς, εμείς την πολυμερή συνεργασία και το γεγονό δηλαδή ότι υπάρχουν εδώ και άλλοι ομιλητέ οι οποίοι ακριβώ συμμετέχουν σε αυτό τον πολυμερή διάλογο. την περασμένη εβδομάδα ε, στην ε, μεγάλη πολυμερή συνάντηση για τα συμβούλια του ε, παγκόσμιου μέλλοντος με έξπατς και διάφορους άλλους ειδικούς σε διάφορα θέματα τα ζητήματα εμπορίου που μας απασχόλησαν ήταν το πώς θα μπορέσει η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη να καταστεί να έχει λιγότερους αποκλεισμούς και το πώς μπορούν να καταρριφθούν μύθοι έτσι ώστε όλες οι κοινότητες να μπορέσουν να συνεισφέρουν πιο επικοδομητικά στις ε, στα ωφέλη που μπορεί να αποφέρει το εμπόριο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο πολυμερή διάλογο μπορεί να διαμορφώσει καλύτερα την εθνική πολιτική έτσι ώστε να αποσβαίνει του κραδασμού αλλά και να υποστηρίζει τι μεταβάσει που θα πρέπει να γίνουν στι εθνικέ οικονομίε σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλά για να επιτύχει κάτι τέτοιο, η εθνική εμπορική πολιτική έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα περιθώρια άσκηση πολιτική για να βρίσκονται τοπικέ λύσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει πολυμερή εμπορική ε, ε, ε, συνεργασία έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολιτικέ οι οποίε θα υπονομεύουν τι γειτονικέ ε, χώρε οι πολυμερείς λοιπόν διάλογος και η συνεργασία είναι ε, πολύ σημαντικές ε, σε ό,τι αφορά και την, ε, τη δουλειά του φόρουμ σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, κατά τις τελευταίους 18 μήνες έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από διαλόγους πολυμερείς σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να ενθαρρύνουμε και τις, τις άμεσε επενδύσει, τι ξένε επενδύσει, ώστε να υποστηρίζουν τι τοπικέ ε, ε, κοινότητε. Και επίση έχουμε μια παγκόσμια συμμαχία σε ό,τι αφορά την ε, διευκόλυνση του εμπορίου. Ω ένα τρίτο παράδειγμα είναι μια πλατφόρμα σε ό,τι αφορά την παγκόσμια αξία που έχουμε δημιουργήσει, προκειμένου να διαρευνούμε καλύτερα τι καινοτομίε που μπορούν να υπάρξουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να είναι πιο δίκαια τα ωφέλη του παγκόσμιου εμπορίου. Επίση θεωρούμε πω η μεγαλύτερη διαταραχή που μπορεί να προκύψει για το εμπόριο στο μέλλον είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι λοιπόν η εμπορική κοινότητα στο πλαίσιο του φόρουμ ε, εξετάζει πολύ ε, στενά ζητήματα του ψηφιακού εμπορίου αλλά και από το ηλεκτρονικό εμπόριο ως και τις διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε εδώ προσπαθούμε να εστιάσουμε σε τέσσερι κύριου τομεί στο πλαίσιο των εργασιών του φόρουμ. Καταρχήν, εξετάζουμε τι βιώσιμε τις βιώσιμες επενδύσει, δηλαδή πώ μπορούμε να έχουμε τον, ε, ένα καλύτερο μηχανισμό διευκόλυνση των επενδύσεων. Από εκεί και μετά εξετάζουμε τη ε, διευκόλυνση του εμπορίου, δηλαδή πώ μπορούμε να έχουμε καλύτερε διασυνοριακέ ροέ ε, δεδομένων και καλύτερη άσκηση σχετικών τοπικών πολιτικών. Επίση, εξετάζουμε την διευκόλυνση του εμπορίου, για παράδειγμα την ενεργοποίηση τη δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο και από εκεί και μετά σε τέταρτη ένα τέταρτο τομέα είναι οι πολιτείε και οι πρακτικέ στο πλαίσιο τη παγκόσμια ε, αλυσίδα αξία, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε κι εσεί, ε, Πρόεδρε. Και προσπαθούμε λοιπόν εδώ να συνεισφέρουμε μαζί με του ε, συναρμόδιου φορεί. Και επίση υπάρχει και ένα, μια πέμπτη πτυχή, δηλαδή αυτή των think tank, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το διεθνέ εμπόριο και τι επενδύσει, όπου εστιάζουμε στο πόσο μπορούμε να επιτείνουμε και να, και αναθεωρήσουμε τι παγκόσμιε επενδύσει, αλλά επίση διερευνούμε και σενάρια και εναλλακτικέ σε ό,τι αφορά το μέλλον του εμπορίου και των επενδύσεων. Όπως σας ανέφερα, είμαστε πεπισμένοι ότι έχει αξία ο ε, πολυμερής διάλογος και αναφέρω εδώ ε, δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχήν έχουμε την πρωτοβουλία του E15 σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ε, όπου είχαμε τη συμμετοχή 400 ε, εμπειρογνωμών και συντάχθηκαν 250 διαφορετικά έγγραφα που αγγίζουν διάφορα θέματα σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, τη καινοτομία, τη διανοτική ιδιοκτησία, τι υπηρεσίε. Ενώ ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η Παγκόσμια Συμμαχία σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση εμπορίου και η οποία έχει εργαστεί καταρχήν στην Κολομβία, δηλαδή σε κάθε ξεχωριστή χώρα όπου γίνεται λαμβάνει χώρα ένα ε, σύστημα ελέγχου των σχετικών επενδύσεων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, εδώ συγκεκριμένα τα τρόφιμα, ενώ στο Μαρόκο είχαμε μια αντίστοιχη ε, διαδικασία σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση των εμπορικών ροών στι λιμένε. Σε αυτήν εδώ τώρα τη διαφάνεια βλέπετε το ε, τους διάφορους ε, συμμετέχοντες εφορείς και βλέπουμε κάποιου εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό τομέα, από τι κρατικέ ε, οργανώσει, από όλε τι υπήρου του κόσμου. Έχουμε και μια σειρά από επιχειρήσει που μα χρηματοδοτούν άμεσα, αλλά και για παράδειγμα το Ομοσπονδιακό της, Υπουργείο της, Αρμόδιο Υπουργείο τη Γερμανίας, αλλά και από, την, από τον Καναδά. Έχουμε υποστήριξη όπω και από τι κάτω χώρε και από την Αυστραλία σε επίπεδο παντοκυβερνητικό. Τώρα, επιτρέψτε μου να σα πω με πιο όρο, όρος ε, ποιε είναι οι σκέψει που κάνουμε σε ό,τι αφορά τρει κυρίου τομεί. Ε, καταρχήν, ε, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό εμπόριο. Οι γλίγορε τεχνολογικέ αλλαγέ επιβάλλουν ακριβώ την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και βέβαια δημιουργούν και κάποιε υποσχέσει σε ό,τι αφορά την, το, το, τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Και βέβαια το ηλεκτρονικό εμπόριο από τι επιχειρήσει προ του ε, ε, καταναλωτέ ε, έχει επεκταθεί ταχύτατα με περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια το 2016. Και οι ηλεκτρονικέ πληρωμέ και μέσω κινητών συσκευών έχουν μεταμορφώσει το εμπόριο, ενώ οι ροέ δεδομένων δημιουργούν ακόμα περισσότερα καινοτόμα μοντέλα, δημιουργώντα περισσότερα από 2,8 3 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ΑΕΠ παγκοσμίω αλλά δεν ε, έχει αποβεί προ όφελο όλων αυτή η ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το 2% μόνο αφορά στι αφρικανικέ επιχειρήσει ό,τι αφορά το διασυναρικό ηλεκτρονικό εμπόριο. 75% των πολιτών δεν διαθέτουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Ενώ ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο ε, εξετάζουμε είναι οι παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής αξίας. Ε, γιατί βέβαια το ίμιση αυτών των αλυσίδων αποτελούνται από τους ε, διάμεσους αν θέλετε παραγωγούς. Ε, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να ε, διαδώσουμε περισσότερες βέλτιστες πρακτικές αλλά να επιτρέψουμε και στις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετέσχουν στο, στην παγκόσμια αυτή αλυσίδα παραγωγής αξίας. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, ειδικότερα στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική, δεν συμμετέχουν σε αυτά τα διεθνή αν θέλετε δίκτυα παραγωγής αξίας. Στις αναπτυγμένες οικονομίες οι εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν καρποθεί πολλά Ενώ η ανησυχία σε ό,τι αφορά ε, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αρμπιτράζ, ενώ και αλλαγέ σε ό,τι αφορά ε, την ανάπτυξη, ε, τι αναπτυξιακέ πολιτικέ έχουν δημιουργήσει μια αρνητική αντίδραση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά ε, τι παγκόσμιε αλυσίδε αξία. είναι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 ε, το που ε, κινούμαστε τώρα προς το μέλλον. Ε, καθώς υπάρχει ένα και περισσότερες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, ε παγκοσμιοποίηση, οι προοπτικές σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο είναι όλο και πιο ανετικές. από την δηλαδή εφαρμογή, εσκεμμένη εφαρμογή κάποιων εμποδίων στο εμπόριο που δημιουργούν διακρίσεις, όπως και η δημιουργία κάποιων συστημάτων που βασίζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες και όσοι σε γενικούς δημιουργούν ένα πιο δύσκολο περιβάλλον σε ό,τι αφορά την άσκηση εμπορικής πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν τρία διαφορετικά σενάρια κατά τη δική μα άποψη από, για το 2017-2020. Το καλό σενάριο είναι ότι ε, τα, ε, η, οι αλλαγέ στην ατζέντα θα παραμένουν εθνικέ, δηλαδή θα υπάρξουν επενδύσει σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τι ε, επαγγελματικέ δεξιότητε αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή των εργαζομένων στι αλλαγέ στην ε, αγορά εργασία. Ε, τώρα, ένα δεύτερο σενάριο είναι το κακό σενάριο. Αυτό θα χαρακτηριζόταν από ανειδική ρητορική αλλά και μονομερή προσεγγίσεις στο εμπορίο. Δηλαδή σε εθνικό επίπεδο θα βλέπαμε ε, συχνή χρήση εργαλείων όπως για παράδειγμα φορολογικέ ε, συμφωνίες ή ε, ε, πολιτική ανταγωνισμού αλλά και ε, κάποια ε, μέσα άσκηση εμπορική πολιτική όπω για παράδειγμα καθεστώτα για τι ρήτρε διασφάλιση των εισαγωγών, μέτρα αντι-dumping, αντισταθμητική διδασμή και ούτω καθεξής. Το τρίτο σενάριο είναι το εξαιρετικά κακό το οποίο θα περιοριζόταν ουσιαστικά σε εμπορικού πολέμου μεταξύ διαφορετικών χωρών και το οποίο θα στόχευε σε συγκεκριμένε επιχειρήσει για παράδειγμα μέσω χειραγώγηση νομισμάτων ή μέσω για παράδειγμα δημιουργίου δημιουργία θέσεων ε, εργασία σε άλλε χώρε, offshore. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα δημιουργήσει και σε αποσάθρωση των γενικών διεθνών θεσμικών οργάνων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια ε, υπεύθυνη άσκηση πολιτική ε, εμπορική και επενδύσεων. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά δικότερα την περίπτωση της Αφρικής, θα πρέπει να καταστήσουμε την ε, πλούσια Αφρική, πλούσια και για τους πολίτες της. Ε, δηλαδή θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε με έναν τρόπο ότι αυτές οι πόροι της Αφρικής θα χρησιμοποιηθούν και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι Αφρικανοί πολίτες. Δηλαδή θα πρέπει ε, αυτέ οι προκλήσει να αντιμετωπιστούν, ε, που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα οι Αφρικανοί πολίτε, για παράδειγμα η ένδυα και η ανισότητα, οι περιφερειακέ πρωτοβουλίε ε, δίνουν τη δυνατότητα για την διεύρυνση του εμπορίου σε ολόκληρη την Αφρική και εδώ θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή τη ε, για τι διαπραγματεύσει οι οποίε συνεχίζονται με την ε, γραμματεία του ε, CFTA στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Αφρικανική Ένωση. Αλλά χρειάζονται να γίνουν ε, και άλλες πρωτοβουλίες από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Επίσης υπήρξε και μια περιφερειακή πρόσφατη πρωτοβουλία από το, από το Global Service Community του Forum που λέγεται hashtag Open Africa, το οποίο περιλαμβάνει την περιήγηση στην Αφρική και, την, και διάφορες συναντήσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή αντίληψη ω προς το τι σημαίνει μια ε, Αφρική. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί ε, να ε, διασκεδάσει του φόβου σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση και το τι αυτό σημαίνει για τι δεξιότητε και τι ε, απασχολήσει. Τώρα σε, σε παγκόσμιο επίπεδο η επίπτωση τη μείωση των τιμών κακάο στην ακτή του Ελεφαντοστού και στην Κάνα, αλλά για παράδειγμα και η διαμαρτυρία σε ό,τι αφορά τη χρήση παιδική εργασία στην αλυσίδε παραγωγή κοβαλτίου που χρησιμοποιείται και στα αυτοκίνητα στην Δημοκρατία του Κογκό υπογραμμίζουν το ότι θα πρέπει να υπάρξουν, υπάρξουν προκλήσει και θα πρέπει πρέπει να δοθούν παγκόσμιες απαντήσεις σε τέτοιου είδους ακόμα και περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, πολλές λοιπόν προκλήσεις και τέλος ο κύριος Ρίτσαρτ Κόζουλ Ράιτ από την UNSTAD που θα εξετάσει τα ζητήματα αυτά κυρίως από την οπτική γωνία των απτυσσόμενων χωρών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ στην Επιτροπή για την ε, πρόσκληση το θέμα, το εμπόριο για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης όταν ε, ζητάμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι, εν μέρη μπορεί το εμπόριο να διαμορφώσει την ε, παγκοσμιοποίηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα παλιό ερώτημα των οικονομολόγων. Οι οικονομίες ποτέ δεν συμφώνησαν σε μια ε, κοινή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο η επιρροή του εμπορίου και κυρίως της εμπορικής πολιτικής εξαρτάται πάντα από διεθνείς δυνάμεις και από ε, τοπικές περιστάσεις και ε, περιορισμούς σε διάφορα επίπεδα. Είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον μέχρι το 1970 ήταν λογικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες να ε, θέλουν να ενταχθούν στην παγκόσμια εμπορική πολιτική. ο δεσμός με τις επενδύσεις έπαιξε σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες της Ιαπωνίας, της Νότιας ε, Κορέας, της ε, Κίνας μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ήταν απαραίτητη μια ενεργή υποστήριξη της εμπορικής πολιτικής πέρα από τα εμπορικά μέτρα. Σήμερα όμως ο κόσμος είναι διαφορετικός. Έχει έχει αναπτυχθεί η παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν σημαντικέ ροές κεφαλαίων και ισχυρές δυνάμεις ε, επικρατούν στην ε, περιφερειακή και παγκόσμια ολοκλήρωση. Τέλος, δεν έχει υποστηριχτεί οι παραγωγικές ε, επενδύσεις ε, επιπτώσεις είναι οι διευρυμένες ανισότητες, η μειωμένη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα και το εμπόριο ε, εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από την, ε, τα αυξημένα επίπεδα του χρέους και αυτό εξηγεί πολλές από τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Από αυτή την άποψη μπορούμε να επαναφέρουμε μια ισορροπία εφαρμόζοντας κάποιους κανόνες, κάποιους, κάποια μέτρα διευκόλυνσης. Αυτό πιστεύουν κάποιοι. Θα ήταν όμως ε, ε, αφελές να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Και το να πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο θα ήταν μια ε, ε επικίνδυνη απάτη, όπως είπε ο Πολ Κρούγμαν, Όλοι πιστεύουμε ότι η επιμονή του Άνταμ Σμιθ για την, το ελεύθερο εμπόριο είναι μια ουτοπία και μια προσεκτική προσέγγιση ε, είναι απαραίτητη. Υπάρχουν όμως τέσσερα ε, ζηματικά ζητήματα. Είναι ε, πλουστευτική, είναι υπερβολική και ε, συγκεχημένη. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι αν θεωρήσουμε ότι το, ανταγωνιστικό το συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να λειτουργήσει για όλους, τότε τα, ε, οι επιπτώσεις ε, είναι, δεν είναι οι επιθυμητές. Αυτό παρατηρήθηκε σε προ, ε, προηγούμενες δεκαετίες, στη δεκαετία του 70, του 80 και γι' αυτό ε, το λόγο το δεκαετία του 90 ο Πολ Κρούγκμαν απέριπτε κάποιες σχετικές αρχές. Σε αυτό το κόσμο το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικά ε, αποτελέσματα αλλά και σε ε, πόλωση της εμπορικής πολιτικής. Πολλοί συμμερίζονται αυτή την ε, άποψη. Είναι υπερβολικό και θα παραθέσω τον Πολ Κρούγκμαν ότι βασίζεται σε λανθασμένους ε, ισχυρισμούς, υπερβολές ε, σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ελευθέρωσης του εμπορίου ε, με βάση ό,τι προβλήπων τα σημερινά οικονομικά μοντέλα. Δεν είναι κάτι τέτοιο ειλικρινές, γιατί μια τέτοια προσέγγιση έχει τη τάση να οδηγεί σε μια λυπή ε, αξιοπιστία ε, και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στην εμπορική πολιτική. Παραδείγματα η Κίνα, η ΙΠΑ, και η συζητή σχετικά με τη Συμφωνία Ναύτα και η σύγχυση. Γιατί, Γιατί δεν, συνεργα... Ε, δεν ανταγωνίζονται οι ε, χώρες, ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν αντιστοιχούν στις χώρες. Το μέγεθος ε, μετράει στο κόσμο του εμπορίου όταν συγκρίνουμε επιχειρήσεις και κυρίως στο διεθνές εμπόριο όπου ε, επικρατούν, έχουν ηγετική θέση οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, μιας χώρας αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του παγκόσμιου εμπορίου. Άρα το ερώτημα είναι πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις θα διαμορφώσουν ε, την παγκοσμιοποίηση και κυρίως πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν ε, στα πλαίσια του, ε, των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων και μπορούμε να δώσουμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι θα, απαντήσουν, θα πούν η απάντηση είναι η καινοτομία, άλλοι με βάση την ε, υλικοτεχνική υποστήριξη της αλυσίδας αξιών. Άλλοι θα απαντήσουν, θα πούν ότι η απάντηση είναι μια επιθετική προσέγγιση. Η απάντηση συνήθως είναι ότι πρέπει να ε, δώσουμε στοιχεία και των τριών αυτών απαντήσεων. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στην επιθετική προσέγγιση των ε, επιχειρήσεων γιατί αυτή η πτυχή έχει αγνοηθεί στις συζητήσεις σχετικά με την παγκοσμιοποίηση και υπάρχουν τρία στοιχεία που βρίσκω στο επίκεντρο των συζητήσεων των οικονομολόγων σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι συνήθως έχουν βραχυπρόθεσμη προσέγγιση μεγάλες επιχειρήσεις και στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Οι παραγωγικές επενδύσεις Πέφτουν όμω, μιας και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κέρδη του για να εξαγοράσουν μερίδια και για να κατανείμουν ε, τα ε, περιουσιακά τους στοιχεία σε ε, φορολογικούς παραδείσους. Τέτοιες επιχειρήσεις συνήθως τον ανταγωνισμό και στις ε, ε, αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. και σε πολλούς τομείς ε, έχουμε όλο ένα και περισσότερες ε, μελέτες σχετικά με τα, τους τεράστιους όγκους κερδών κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων αύξηση των τιμών, αύξηση των κερδών ε, σε πολύ υψηλά επίπεδα και Συνήθω επιχειρήσει την να παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοτική ε, ε, ιδιοκτησία και διάφορες αρχές που χρησιμοποιούν, παραβιάζονται προκειμένου να ε, παραβιαστούν, να αυξηθούν τα κέρδη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των παραγωγικών επενδύσεων. Ενώ πολλές ε, αναπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, ε, αυτές οι τάσεις παρατηρούνται και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και κλείνοντας θα έλεγα ότι βρήκαμε απαντήσεις από το ε, Πανεπιστήμιο του Σικάγο σχετικά με τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Άρχισαν να μιλάνε για ένα ε, φαύλο κύκλο όταν περιγράφουμε τη σχέση ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολιτικές διαδικασίες. Γιατί φαίνεται να ε, λειτουργούν όπως το 16ο αιώνα και όχι όπως θα έπρεπε στη σύγχρονη εποχή. Ευχαριστώ πολύ. Okay, μήνυμα. Πριν από 150 χρόνια ε, δημοσιεύθηκε το κεφάλαιο. Οι συναδέλφοι μου έχουν το λόγο για ένα λεπτό. Πρώτον, ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ πως το ερώτημα δεν έχει τεθεί με το σωστό τρόπο, δηλαδή αν αυτή η στρατηγική ε, για το εμπόριο για όλους θα συνδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο ή όχι. Φυσικά και θα συνδιαμορφώσει, αλλά με ποιον τρόπο αυτό είναι το ερώτημα. Ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να βασιζόμαστε στο αόρατο χέρι της αγοράς, έτσι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυτό το αόρατο χέρι δεν υπάρχει. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους στόχους της δυόμισης ανάπτυξης των ε, Ηνωμένων Εθνών, ε, τι θα πρέπει να πούμε, ότι αν θέλουμε να υπάρξει μια θετική συμβολή, τότε θα πρέπει να συνάδει με αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, οποιαδήποτε ε, στρατηγική διαχαράξουμε θα πρέπει να είναι εφαρμοστές στην πράξη γιατί συνδέει μεταξύ τους δύο πράγματα. Μία, ε, ελεύθερη άσκηση εμπορικής πολιτικής σε πολυμερές επίπεδο και από την άλλη περιφερειακή ε, διάσταση αυτής της πολιτικής αλλά και λήψη υπόψη άλλων παραμέτρων για παράδειγμα σε ό,τι αφορά εργασιακές σχέσεις αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, εάν σκεφτούμε λίγο παραπένω, παραπάνω ε, δεν μπορούμε να επιμείνουμε μόνο στη σύναψη ε, συμφωνιών ελεύθερου αμπορίου. Θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλε πολιτικέ. Αλλιώ θα ήμασταν πολύ αφελεί. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την άσκηση εμπορική πολιτική ε, σε σχέση με την Κίνα. Και βλέπουμε πόσο συγκεκριμένα ασκεί πολιτική η ε, Κίνα, για παράδειγμα, της, ε, ε, την επενδυτική της πολιτική, τις επενδυτικές της δραστηριότητες με πολύ επιτυχημένο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν με αντίστοιχο τρόπο και εμείς θα πρέπει να χαράξουμε αντίστοιχες συνοδευτικές πολιτικές πέρα από την εμπορική. Και Ίσως θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες σκέψεις με στους επόμενους μήνες και χρόνια. Για παράδειγμα υπάρχουν ε, ε, οι δυνατότητες σύναψης οικονομικών, ε, συμφωνίων οικονομικής συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες. Αλλά ενώ εκεί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα, ένα κακό παράδειγμα είναι οι συμφωνίε στο πλαίσιο τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, όπου είναι μάλλον μόνο ελεύθερο εμπορίο συμφωνίε και τίποτε άλλο. Κυρία Ροντρίγκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου του ομιλητέ. Πολύ σύντομα. Ε, θα κάνω κάποιες ερωτήσει προς τον κύριο Βόλφα για την παγκοσμιοποίηση. Είναι σημαντικό να βάλουμε τη διάσταση του φύλου στην εμπορική πολιτική. Ε, ποια θα είναι η επίπτωση του ΠΟΕ ούτως ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Προς τον κύριο Κόσουλ Ράιτ. Είσαστε οικονομολόγος και εγώ είμαι οικονομολόγος αλλά δεν πρόκειται να πάρω ποτέ βραβείο Νόμπελ. Ε, ε, κυρία Κάνσε, επίσης, γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα της στόχιας σε χώρες λιγοτών Και αν δεν κατάλαβα λάθος, μα ζητάτε μια παγκοσμιοποίηση που θα βοηθάει την Αφρική για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο εμπόριο. Μου το σχολιάστε λίγα και αυτό. Φυσικά η παγκοσμιοποίηση έχει μεγάλη σημασία στην εμπορική πολιτική, γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ και τα συζητάμε αλλά έχει και τεράστια πολιτική στο πώς ε, διανέμονται τα κέρδη από τις εθνικές πολιτικές. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν, ε, στην πραγματικότητα γίνεται μία, ε, ένας ανταγωνισμός για να προσελκύσουν πολυεθνικές που θα πληρώνουν όλο και λιγότερους φόρους. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια δραματική κατάσταση. Γιατί αυτέ οι χώρε είναι ακριβώ αυτέ οι χώρε που χρειάζονται περισσότερο φορολογικά έσοδα για να ε, χρηματοδοτήσουν την ε, υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Στα διεθνή φόρουμ τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε που το χρειάζονται περισσότερο. Χρειάζονται περισσότερα αυτά τα έσοδα από τι πολυεθνικέ, οι οποίε δεν τα πληρώνουν. Ευχαριστώ. Μία άμεση ερώτηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας διαγραφήθηκε από τον Ρίτσαρντ, μια υπερπαγκοσμιοποίηση που δημιουργεί σε μια σε υπερβολικά χρηματοδοτικά ε, κινήσεις, ας πούμε, σε ανισότητες βορρά-βορρά και νότου-νότου. Ε, η υπερσυγκέντρωση ε, δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις, πούμε, του ανταγωνισμού. Εκεί υπάρχουν από τη μία οι οποίοι ε, είναι υπέρ της, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και από την άλλη άλλοι που είναι υπέρ του εμπορίου. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και ποιες, ποια είναι τα, οι προϋποθέσεις μία εμπορική συμφωνία. Όταν διαβάζουμε την έκθεση της UNCTAD για το εμπόριο και την ανάπτυξη βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το εμπόριο που έχει σημασία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις ε, που πρέπει να προηγηθούν των εμπορικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. Έχω διάφορες ερωτήσεις που δεν νομίζω ότι έχουν ε, απαντηθεί. Το, εμπόριο, το ελεύθερο εμπόριο είναι σαφώς ε, θετικό πράγμα. Πάντα, παλιά το πίστευα, τώρα έχω αμφιβολίες. Το ελεύθερο εμπόριο είναι καλό και το περισσότερο ελεύθερο εμπόριο είναι ακόμα καλύτερο. Το να ε, υπάρχουν περισσότερες θέσεις ε, απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι καλό πράγμα. Δεν αναφέρθηκε από ό,τι ήταν παρά μόνο έτσι γενικόλογα, το θέμα των υπηρεσιών. Σε ποιο βαθμό ο ΠΟΕ είναι αποτελεσματικός στο να καλύπτει τις υπηρεσίες. Ο κύριος Βόλφ ε, είναι εντυπωσιακό, κοίταξα λιγάκι το βιογραφικό του ενώ μιλούσε. Ε, είπε ότι αν το τι είχε περάσει, θα υπήρχε ένα, μια παγκόσμια δομή ρυθμιστικού χαρακτήρα. Η άποψη πολλών μας, όχι μόνο ε, δεξιών και αριστερών, είναι ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και, τις και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα είχαν να κάνει πάρα πολύ καλό λόμπι για να δυσκολέψουν τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν είχε περούσε το TTIP. Ε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι σχετικό και τέλος. Σε πέντε λεπτομέρεια. Σε πέντε δευτερόλεπτα. Ήσασταν πάρα πολύ εύγλωτοι όλοι σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως είναι μια, ένα μπλοκ υπέρ του προστατευτισμού. Ε, όσοι είσαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, δεν θα πρέπει να είσαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των κανονισμών. Θέλω να δω τι θα κάνει η Βρετανία όταν φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, θα το δείτε. Συγγνώμη, αλλά εγώ πρέπει να φύγω σε λίγο, γιατί έχω ένα τρένο που πρέπει να μην χάσω. Um, ένα ερώτημα και από τη δική μου πλευρά. Άκουσα πολλά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε και σε ένα είδος, για παράδειγμα, κανονισμού, ε, antitrust Νομίζω ήδη στην περίοδο Ροκεφέλερ είχε γίνει μια τέτοια πρόταση. Κύριο Κόζουλ Ράιτ, ναι, ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να πάρω ένα τρένο για να απαντήσω κατευθείαν σε αυτό το τελευταίο ερώτημα. Ναι, το αντιτράστ, δηλαδή η πολιτική αντιτράστ, ε, έχει τεθεί και πάλι επιτάπητο ε, πρόσφατα στι ΗΠΑ ε, και αν το σκεφτεί κανεί, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια αρχή, παγκόσμια αρχή σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Αποκλείται να υπάρξει στο έγκυο αλλά υπάρχει μια. είναι λογικό το να υπήρχε μια τέτοια αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη ε, πολιτική σε σχέση με τα όσα είπα. Ναι, εγώ είμαι ε, μεγάλος οπαδός αυτού το οποίο ε, ονόμασε ε, κάποιος μελετητής ε, των ΗΠΑ ως ρεαλιστικό πειραματισμό. Ε, εγώ θα αναφερνόμουν δηλαδή περισσότερο στην εμπειρία στην Ανατολική Ασία μετά τον δεύτερο α, α, παγκόσμιο πόλεμο. Πάντως αυτό που χρειαζόμαστε σε σχέση με αυτόν τον ρεαλιστικό πειραματισμό είναι τα απαραίτητα περιθώρια άσκηση πολιτική για όλε τι χώρε έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τι επιμέρου συμφωνίε, τι συγκεκριμένε προκλήσει, τι οποίε αντιμετωπίζουν και δυστυχώ αυτό δεν ισχύει στο πλαίσιο των περισσότερων συμφωνιών οι οποίες ε, ε, έδωσαν υπερβολική έμφαση στην περικοπή των διαφορών εναλλακτικών που έχουν στη διάθεσή του οι αναπτυσσόμενε χώρε και οι οποίε ε, έχουν καταδείξει την αξία του στο μέλλον. Δεύτερον, δεν μπορεί κανεί να ασκήσει εμπορική πολιτική σε έναν κόσμο ε, μη σταθερών και αβέβαιων ε, χρηματοοικονομικών ροών και σχετική αστάθεια. Αυτό δηλαδή είναι και το συμπέρασμα που προέκυψε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν μπορεί κανεί επίση να ασκήσει εμπορική πολιτική στο πλαίσιο ε, πολιτικών λιτότητας. Ε, κάτι τέτοιο δηλαδή σίγουρα θα παράξει δύο ε, την αστάθεια και ανισότητα. Και νομίζω πως αυτό βλέπουμε και στην πράξη να συμβαίνει κατά τα τελευταία 5-6 έτη. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε εμπορική πολιτική σε ένα κόσμο λιτότητας. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια μακροοικονομική πολιτική η οποία θα αντισταθμίζει λίγο αυτό τον αντίκτυπο. Και από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά την Αφρική, ναι, η Αφρική κατά τι τελευταίε τρει υπήρου ε, προβαίνει στι περισσότερε εμπορικέ αλλαγέ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ήπειρο ε, κατά ε, του τελευταίες τρεις αιώνες αλλά δεν το κάνει με το σωστό τρόπο γιατί ακριβώ προβαίνει στην εμπορία κομμωδίτη χωρί να έχει δημιουργήσει μια βιομηχανική βάση χωρί μια σοβαρή και διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση δεν μπορεί να προβεί σε κατάλληλε εμπορικέ συναλλαγέ και δεν νομίζουμε ότι αυτή η βάση θα δημιουργηθεί μέσω απλώ και μόνο του ανοίγματο των αγορών αυτών στις διεθνείς συνεργασίε και στο ελεύθερο εμπόριο. Θα δημιουργηθεί αυτή η βάση μέχρι της αυστηρής ανάπτυξης των καταλήλων ε, ικανοτήτων και των, δομών, και των επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορέσουν να είναι κεντροφόρε σε λόγω χώρες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, οπότε επειδή και ο κύριος Βόλτ θα πρέπει να αποχωρήσει, θα, θα του δώσω το λόγο για δύο λεπτά και μετά θα ακούσουμε και κάποιες ακόμα παρεμβάσεις από κάποια ακόμα μέλη. Οι διαπραγματευτές σε ό,τι αφορά εμπορικά ζητήματα ασχολούνται με πρακτικά θέματα. Ε, και ένα από τα ζητήματα που τέθηκε στην ε, μερίσα διάταξη τη Υπουργική Διάδευση ε, που θα λάβει χώρα σε τρει εβδομάδε στον Μπουένο Άρε είναι η ενισχύση στον χώρο τη αλληλεία. Δεν πρόκειται εδώ για ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί διστάμενε απόψει ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσει για τον Νότο. Ε, δηλαδή και οικονομικέ επιπτώσει, αλλά και ε, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο Κρούγκμαν για κάτι τέτοιο, ή αν ο Κέιν, για παράδειγμα, φοβόνταν για τα ψάρια ή όχι, αλλά σίγουρα εμεί φοβόμαστε. Και υπάρχουν τεράστιε ενισχύσει οι οποίε ε, δίνονται τελικά σε κάποιε αλληλευτικέ επιχειρήσει, των οποίων τα αλληλευτικά σκάφη πραγματικά αδειάζουν ε, τις, ε, τις ε, θάλασσες και έχουν πολύ σημαντικές αντικές οικονομικές συνέπειες για άλλες χώρες. τώρα, εγώ είμαι πρόεδρος ε, μιας ομοσπονδίας βάμακο που βρίσκονται σε πολύ φτωχές χώρες της Αφρικής, Τσάντ, Μαλή, Μπενίν και Μπουρκίνα Φάσο και όλοι ε, έχουν δεσμευτεί στο να παράσχουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους ε, παραγωγούς αυτούς, ε, σε αυτές τις εξαιρετικά φτωχές χώρες. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή βάμβακος, είτε μιλάμε για παραγωγούς ή για χώρες παραγωγούς βαμβακιού, είτε για χώρες καταναλωτές, όλες, όσες συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία υποστηρίζουν εδώ αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Επίσης σε ό,τι αφορά την ψηφιακή επανάσταση και πάλι εδώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση εδώ. Ε, Βορρανότου, για παράδειγμα το ε, Πακιστάν, η Νιγηρία ε, και άλλοι θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη έμφαση σε αυτή τη διάσταση σε ό,τι αφορά το μέλλον του εμπορίου και αναφέρθηκε για παράδειγμα από την πλευρά του Πακιστάν ότι από τη μηδενική του συμμετοχή του στο διαδίκτυο τώρα ο μισό ενήλικο πληθυσμό, 47 εκατομμύρια άτομα ε, ε, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό, ότι είτε είμαστε στις ΗΠΑ είτε είμαστε σε αναπτυσσόμενες χώρε, υπάρχει μια ε, ευκαιρία συμμετοχής στο διεθνέ εμπόριο. Και δεν είναι όλες μεγάλε μεγάλες πολυεθνικέ επιχειρήσεις κακές. Το eBay και άλλες τέτοιες πλατφόρμες είναι πλατφόρμες για την ε, παγκόσμια ε, διάθεση στην αγορά των διαφόρων προϊόντων από διάφορες χώρες. Ε. Και επίση δημιουργεί και περισσότερε ευκαιρίε αυτό το ελεύθερο εμπόριο και για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Γιατί πολλέ μικροεπιχειρήσει ακριβώ τρέχουν από γυναίκε. Βρίσκονται από την διάθεση γυναικών. Οπότε προφανώ χρειαζόμαστε πολύ χρόνο. Και για παράδειγμα η αρχική συμφωνία σε ό,τι αφορά τον ΕΠΟ προβλεπόταν να έχει συναυθεί το 1990, τελικά ε, συναυθεί το, το 1994, οπότε πραγματικά όταν εδώ συζητάμε για ε, παγκόσμιο εμπόριο, συζητάμε για ρεαλιστικά ε, ε, προβλήματα, για προβλήματα πρόσβαση στη διεθνή αγορά και ό,τι καθεξή. Οπότε σα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση, στο συγγνώμη που θα πρέπει να αποχωρήσω και πραγματικά σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχα να παρακολουθήσω και τις παρεμβάσει των υπολείπων και των ομιλητών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε θα είμαστε σε επαφή και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Πολλές άλλες φορές. Κυρία Κάντσα. Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια. Θα εστιάσω στο θέμα του πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε την ε, παγκοσμιοποίηση για να επεκταθεί το, και να συμμετάσχει περισσότερο η Αφρική στην, ε, στο εμπόριο. Δύο στατιστικές. Ε, Κάτι που ανέφερε και ένας άλλος ομιλητής. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα στην Αφρική να κάνει περισσότερο εμπόριο. Αν κοιτάξουμε τη βάση για την εκβιομηχάνηση, με βάση την Αφρικανική Τράπεζα, ε, η, η... η Αφρική εξάγει βιομηχανικά αγαθά λιγότερο από το 1% σε σχέση με το 16% της ε, Ανατολικής Ασίας. Ε, πρέπει να, ε, να ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό του 1%. Και χρειάζονται επίση και υποδομέ, μεταφορέ. Με βάση την Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική του ΟΗΕ, ε, το, το κόστο μεταφορών για τις θύλακε, για τις χώρες που είναι θύλακες και δεν, είναι, έχουν πρόσβαση στην θάλασσα δηλαδή, έχουν υψηλότερε μεταφορέ κατά 70%. Ε, η διασύνδεση τη Αφρική ε, δεν είναι επαρκή. Αν κοιτάξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και πώ μπορούμε να αυξήσουμε τον, το δυναμικό των μικρομεσαίων για να συμμετάσχουν στι περιφερειακέ και παγκόσμιε αλυσίδε αξιών, γιατί υποεκπροσωπούνται συχνά, το θέμα είναι ότι έχουν χαμηλό δυναμικό, δεν ε, είναι στο επίπεδο των παγκόσμιων προ... Προτύπων. Το θέμα είναι ε, όπω η κότα και τα αυγό. Τι περιμένουμε μέχρι να μπορέσουν να αυξήσουν τα, το επίπεδό του για να φτάσουν στο επίπεδο Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι στην Αφρική ε, οι μικρομεσαίες ε, διευθύνονται από γυναίκες, ε, νέους κτλ. Θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις για να καλυφθεί το κενό. Εγώ μιλάω πολύ για τις προκλήσεις της δυσκολίας. Θέλω να είμαι πιο αισιόδοξη. βλέπουμε την Αφρική και κυρίως τη Νέα Αφρική να ασχολείται περισσότερο με την ε, ψηφιακή οικονομία, εκεί όπου υπάρχει διασύνδεση και το πρακτικό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι καθώς η Ευρώπη αναπτύξει, αναπτύσσει το ψηφιακό τη πλαίσιο, να μην ε, υψώσει προστατευτικά τείχη και να διευκολύνει το εμπόριο, ειδικά το ψηφιακό εμπόριο, μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, των Αφρικανών και των Ευρωπαίων. Και τελευταίο και σημαντικό είναι το θέμα των οικονομικών ροών. Ε, είναι σημαντικό πού θα προέλθουν αυτέ οι επενδύσει. Ε, υπήρχε μια ε, μελέτη που έγινε για την παράνομη χρηματοδότηση, μάλλον παράνομες οικονομικές ροές στην Αφρική. Ε, μιλάμε για φορολογική διαφυγή, για το transport pricing. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, σπάσουμε αυτές τις κερκόπορτες, να τις κλείσουμε αυτές τις κερκόπορτες και να βρούμε κάποιους πόρους που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ε, με παραγωγικό τρόπο και να συνεισφέρουν και να συμπληρώσουν τις ε, συμφωνίες ε, ελευθερού εμπορίου. Εγώ είμαι υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης και πιστεύω ότι αν το δούμε από όλες τις σκοπιές τελικά είναι κάτι θετικό η παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Κλείνουμε. Η κυρία Σάιφη, η συγγήτριά μας, θα κάνει τα τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το σύνολο των ε, ομιλητών. Η Ομιλιε ήταν πλούσιε ε, και δείχνουν τι πολυάριθμε τις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα στην εμπορική πολιτική. Το διεθνέ εμπόριο και οι αλληλεπιδράσει του άλλαξαν ε, εν, το βάθρο εδώ και δύο χρόνια. Ε, νέες προκλήσεις και υπάρχει μια ενδιάμεση αναθεώρηση τη στρατηγική μα, απαραίτητη μάλλον για να προσαρμόσουμε τις ε, πράξει μα και να απαντήσουμε στου διάφορου στόχου. Αυτές οι νέες προκλήσεις ε, βασίζονται σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο εξελίχθηκε πρόσφατα και είναι σε συνεχή μετασχηματισμό. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην, ε, στη δημιουργία του παγκόσμιου ε, συστήματος από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Εμπορίου Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σημερινές ε, είπα του Τραμπ δεν θέλουν την πολυμέρεια και δεν θέλουν νέες ε, εμπορικές συμφωνίες, ούτε παγκόσμιους πολυμερείς κανόνες. Ο κύριος Γουλφ τα είπε πολύ ενδιαφέροντα αυτά, με πολύ ενδιαφέρον τρόπο προηγουμένως. Η Ασία παράλληλα ε, γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και θέλει και εκείνη να συνδιαμορφώσει τους διεθνείς κανόνες. Σήμερα παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη εμπορική δύναμη παγκοσμίω, οι προβλέψει βλέπουν ότι μέχρι το 2000, λένε ότι μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μόνο το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ 23,7% ήταν το ποσοστό το 2013. Θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, ούτω ώστε να κρατήσουμε μια δυνατή Ευρώπη ε, που θα παίζει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Οι συζητήσει που είχαμε σήμερα με, τις, ε, με τους διάφορους ομιλητές υπενθύμησαν τις ε, βελτιώσεις που πρέπει να επιφέρουμε κατά την εφαρμογή των συμφωνιών, ούτω ώστε να είναι για όλους και να συνεισφέρουν σε ένα δίκαιο εμπόριο. Από την άλλη, Είμαστε στα πρόθυρα τη 11ης Υπουργικής Διάσκεψης, ε, ακριβώς γι' αυτό ο ΠΟΕ χρειάζεται πολύ περισσότερο παραποτέ την υποστήριξή μα και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μα για να ενισχύσουμε του πολυμερει κανόνε. Τη δεύτερη μέρα της, αυτής της εμπορικής πολιτικής που οργάνωσε η, η Επιτροπή ΙΝΤΑ ήταν πολύ χρήσιμες συζητήσεις και ως εισηγήτρια θα λάβω υπόψη μου πολλά από τα στοιχεία που άκουσα σήμερα. Ευχαριστώ όλους τους προκεκλημένους για τις πολύτιμες συνεισφορές τους. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ε, συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Ε, δεν ολοκληρώνεται εδώ βέβαια αυτή η συζήτηση, αλλά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους και ας μείνουμε σε επαφή. Okay, so, uh, dear colleagues, Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή το σημείο 8 της Μέσας Ένταξης, τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία. Βλέπω πως πολλοί αποχωρούν από την αίθουσα και δεν ε, μπορώ να καταλάβω γιατί. So, ε, point eight. And, ε, Σημείο λοιπόν 8. Ναι, και εδώ να σας διαβάσω δύο ειδήσει, αν θέλετε δύο στοιχεία. Ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι ότι ο κύριος Σατάκουλα θα καταλήψει την Επιτροπή μας. Το καλό νέο είναι ότι θα είναι πλέον ε, μέλος του Ελεκτικού Συναδρίου, οπότε τον συγχαίρουμε για την εκλογή του εκεί. Και ίσως, ποιος ξέρει, να είναι αρμόδιος στο μέλλον. Στο μέλλον για αυτό το σημείο εδώ, για αυτό το ζήτημα, για το οποίο είναι συγητής τώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε έχει το λόγο. So, to... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τη 1η Μαρτίου θα ξεκινήσω στο Λουξεμβούργο, μένουν λοιπόν τρει μήνε και ελπίζω ότι θα έχουμε και άλλε καλέ στιγμέ σε αυτό το διάστημα. Ελπίζω επίση ότι θα μπορέσω να επιτύχω ε, κάτι και στο δικαστήριο σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Και εκεί ο πρόεδρος είναι γερματός. Από γερμανική προεδρία σε γερμανική προεδρία. Φετικά όλα αυτά πάντως. Όπως ε, λέμε, ας ε, περάσουμε στην ουσία. Είναι τρίτη φορά που προτείνεται χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία μετά ε, το 2008. 10 εκατομμύρια θα δοθούν σε 35 εκατομμύρια σε δάνεια και 10 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις. Ε, η χώρα βρίσκεται σε ε, δύσκολη γεωπολιτική θέση, αντιμετωπίζει προκλήσεις και έχει υψηλό δημόσιο χρέος η οικονομία επιβραδύνθηκε επειδή έπεσε το ποσοστό των ε, εξαγών, το ΑΕΠ αυξήθηκε κυρίως χάρη στις επενδύσεις και σε ό,τι αφορά διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία, έχουν επιληθεί πολλά, αλλά και άλλα ε, πρέπει να επιληθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία πρόσφατα σύναψαν μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που συμφάλει στη σταθεροποίηση της οικονομίας της Γεωργίας. Η προτινόμενη χρηματοδότηση ε, είναι ανάλογη και καλύπτει εν μέρη το εφιστάμενο ε, χρηματοδότησης και θα βοηθήσει την οικονομία της Γεωργίας. Ελπίζω η Επιτροπή αυτή να υποστηρίξει αυτή την πρόταση και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι συνεργαζόμαστε στενά και με άλλες επιτροπές και χαίρομαι που μου δίνεται αυτή η δυνατότητα ε, μαζί πήγαμε και στη Γεωργία, επισκεφτήκαμε ε, κάποια μέρη και έχουμε λοιπόν εμπειρία από ε, την πραγματικότητα επιτόπου. Κινούμαστε λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον εισηγητή της Επιτροπής ΑΦΕΤ, τον κύριο Μαμίκινς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ως ε, ε, εισηγητής της ΑΦΕΤ για τη Γεωργία, όπως είπε και ο συνάδελφος, η προηγούμενη εβδομάδα συνήφθη συμφωνία με τη ε, Γεωργία. Φυσικά, για μένα είναι πάντα μεγάλη χαρά να, να συνεργάζουμε το κύριο ε, Τάκουλα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιστήσουμε την προσοχή σε διάφορα ζητήματα που εξετάζουμε κυρίως σε ό,τι αφορά ζητήματα που ενόρχονται συχνά ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων. Το πρώτο, το μνημόνιο συμφωνίας, Ε, όπου ε, ορίζονται οι όροι που πρέπει να τηρηθούν από την ε, δικαιούχο χώρα. Δεύτερον, η αξιολόγηση των προϋποθέσεων για το MFA και τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Και το τρίτο σημείο, τα διδάγματα που αντλήσαμε από τα προηγούμενα MFA. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα δύσκολο χρονοδιάγραμμα εργαζόμαστε στεναρά προκειμένου να ε, σας δώσουμε την απαιτούμενη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Χάνου Τάκουλα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένας από τους πολλούς ευρωβουλευτές που θα προωθήσουν ε, τις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν είναι ο μόνος, συγχαρητήρια όμως. Και ε, καλωσορίζω τον συνάδελφο από την ΑΦΕΤ και συνεισηγητή. Τα βασικά στοιχεία ακούστηκαν. Εμείς από το ΕΛΚ πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ξεκάθαρα ε, για το μνημόνιο συνεννόησης τη ρήτρα αρεσιμότητας, τις προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα MFA. Επίσης παρακολουθούμε την κατάσταση στη Γεωργία και από ό,τι ξέρουμε η εξέλιξη της χώρας είναι καλή. Βεβαίως υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιωθούν ακόμα. Καταρχά το κράτο δικαίου, αναφέρθηκε ήδη συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά και κάποιες αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στην οικονομία. Ε, η μακροοικονομική βοήθεια θα θέλει να αντιμετωπίσει αυτούς τους τομείς. Στην πραγματικότητα συμπληρώνουμε τις προηγούμενες παρεμβάσεις που κάναμε στη Γεωργία και σεβόμαστε την Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωση Γεωργίας. Είδατε ότι υπάρχει και μια αξιολόγηση στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου και η ιδέα ποια είναι, ότι θα πρέπει μέσω της εφαρμογής αυτού του προγράμματος ε, μακροοικονομικής ε, βοήθειας να βελτιώσουμε και την DCFTA Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας, τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου εις βάθος και πλατιά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Ελπίζω να περάσει ε, αμελητή το θέμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ζαραντήλ. Και εμένα με ενδιαφέρει η Γεωργία Ήμουν τον Ιανουάριο και θα ξαναπάω σε δύο εβδομάδε. Ξέρω την κατάσταση από πρώτο χέρι. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι μια χώρα τεράστια σημασία. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να την λάβουμε υπόψη μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικά θα πρέπει να ασχοληθεί με τη Γεωργία. Συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν. Δεν ε, γίνεται για πρώτη φορά που δίνουμε μακροοικονομική βοήθεια στη Γεωργία. Η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες, είναι ευάλωτη, όχι μόνο πολιτικός πώς, αλλά και οικονομικός πώς. Είναι θετικό το ότι φέρνουμε κάποια μέτρα που μπορούν να σταθεροποιήσουν περαιτέρω τη χώρα. Φυσικά μπορούν να βελτιωθούν κάποια πράγματα, να υπάρχει καλύτερη ανατροφοδότηση, καλύτερο feedback ε, για το αποτέλεσμα των δράσεών μας. Μονίμως ζητάμε γραπτές εκθέσεις, το ξέρω, και παρακολούθηση εκ του Ίσως θα πρέπει όμως να καλούμε πιο συχνά την Επιτροπή εδώ για να λογοδοτεί και να μας εξηγεί ποια είναι τα αποτελέσματα των δράσεών μας αλλά γενικά η βοήθεια αυτή είναι θετική και την υποστηρίζει και η ομάδα μου. Φυσικά, ε, και εγώ τον ε, συνάδελφο από την ΑΦΕΤ. Γενικά έχουμε θετική στάση και θα υποστηρίξουμε την κίνηση αυτή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Νέος αιώνας ε, έχει ανατείλει στη σχέση μας με την ΑΦΕΤ. Θαυμάσιο πράγμα αυτή η συμφωνία που κάναμε εγώ και ο πρόεδρος της ΑΦΕΤ. Μέσα αυτό το αγαστό πνεύμα συνεργασίας ελπίζω να, τα, να, συνεχίσουμε. Εμείς το καταψηφίσαμε, το, κείμενο αυτό. δεν θέλουμε να μπει ακόμα μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. προσωπι... προσωπικό σχόλιο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τάκουλα που εξελέγει για το ελεκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω ποια είναι τα πρόσφατα του κύριου Τάκουλα ακριβώς. Πάντως μιλάμε για 45 εκατομμύρια που θα πάνε στην ε, Γεωργία. Και μια και ο κύριο Στάκλο θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο, θα ήθελα να μου πει πώς ε, θα παρακολουθήσουμε την κίνηση αυτών των ποσών. Ρίχνουμε το τσουβάλι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή. Αλλά κανένα δεν έχει καμία εμπιστοσύνη ότι τα λεφτά αυτά θα ξοδευτούν σωστά. Αν πιστεύετε ε, στο σύστημα. Εγώ δεν το πιστεύω βέβαια, αλλά αν πιστεύετε σε αυτό το σύστημα, ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να σε απασχολήσουν είναι να ξοδεύονται σωστά τα λεφτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Λεφτά που δίνουν με το τσουβάλι στη Γεωργία. Τουλάχιστον ξοδεύονται σωστά. Τα λεφτά είναι εδώ για να καλύψουν τις εξωτερικές ε, δανειακές ανάγκες της χώρας. Ακόμα και αν καλύψουν αυτές τις ανάγκες τα λεφτά, θα χρειάζονται άλλα κονδύλια ε, για να τα ξοδέψει όπως θέλει η Γεωργία, έτσι. Δεν θα μας συζητήσω τώρα επί της αρχής. Αλλά πάντως θα ήθελα να μου πει ο κύριος Στάκουλα, μια και θα αναλάβει τη θέση που θα αναλάβει, πώς προτείνεται οι δαπάνες αυτές από τη Γεωργία και τα υπόλοιπα λεφτά που θα δώσουμε στη Γεωργία, να τα παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε το πώς ξοδεύονται, γενικά να τα ειχνηλατούμε. Σημαντική ερώτηση βεβαίως. Και θα, θα συζητάμε αντίστοιχα και όταν φτάσουμε για να δίνουμε μακροοικονομική βοήθεια στη Βρετανία τα ίδια θέματα. Κύριε Τάκουλα, βεβαίως, να απαντήσετε. Ναι, να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ε, σημαντικό να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το πώς δεπανώνται αυτά τα χρήματα και θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον έλεγχο που θα κάνουμε σε σχέση με το που κατευθύνονται τα χρήματα. Κάποιος από την δική σας πλευρά, από τον Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ότι Ε, επιχειρηματολογούσε κάποτε ότι θα μπορούσε ε, να εξοικονομηθούν ε, εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ τα οποία από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κατευθυνθούν στο δημόσιο σύστημα υγεία. με το ίδιο σκεπτικό οι μέθοδοι τις οποίες εφαρμόζουμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ελέγχων ε, θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν και εδώ σε σχέση με το Γεωργείο τους ώστε πράγματι να είναι κατάλληλα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή τώρα θα λάβει το λόγο. Και να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα από τη δική μου πλευρά. σε ό,τι αφορά και μια παρουσίαση που έκανε και το ελεκτικό συνέδριο πριν από μερικέ εβδομάδε. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι οι ρεσιμότητε ε, μόνο σε 5 από τις 15 συνολικά περιπτώσεις ελέγχονται και παρακολουθούνται με τον κατάλληλο τρόπο. Οπότε τι συμβαίνει ε, στην, ε, στη δική ε, από την πλευρά της Επιτροπής. Πράγματι ισχύει αυτό. Ο κύριος κύριε Γκρίζε λοιπόν από την πλευρά της Επιτροπής. Ναι, είμαι γενικό σε ό,τι αφορά τα οικονομικού χαρακτήρα ζητήματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, μακροοικονομική ε, υποστήριξη ή ενίσχυση προ τη Γεωργία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου που ε, υποστήριξαν τη δική μας αυτή πρόταση και προτού απαντήσω τώρα στα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν, επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι ευθύ εξ αρχής. Υπάρχουν δύο μικροπροβλήματα σε ό,τι αφορά το κείμενο της απόφασης ε, το οποίο υποβάλαμε στις 29 Σεπτεμβρίου τα οποία ήδη έχουν αναφερθεί και στο σχέδιο έκθεση ε, του κ. Τάκουλα και για τον οποίο τον ευχαριστούμε. Για την οποία αναφορά τον ευχαριστούμε. Το ένα λοιπόν από αυτά τα προβλήματα ή μάλλον και τα δύο αφορούν το άρθρο 4 ε, δηλαδή την παράληψη εδώ της λέξης του ότι δηλαδή η, ε, αυτή η μακροοικονομική ενίσχυση θα πρέπει να παρέχεται σε δύο δόσεις ε, και στο άρθρο 2 όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ό,τι αφορά την εκταμείευση αυτή τη υποστήριξη ε, ε, με βάση την πλήρωση όλων των αριθμοτήτων. Ε, άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διατύπωση του κειμένου και είμαστε σε φάση τώρα δημοσίευση ενό διορθωτικού ενό προκειμένου ακριβώ αυτά τα δύο συντακτικού χαρακτήρα ζητήματα να έχουν διορθωθεί προκειμένου να έρθει με το σωστό τρόπο από του σύνομοθετέ στο κείμενο. Τώρα, περνώντα στο ίδιο το περιεχόμενο τη πρότασή μα. Όπως αναφέρθηκε από μια σειρά από ε, το γενικότερο πλαίσιο αυτή τη πρόταση είναι το γεγονό ότι η γεωργία ε, παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα εξυπηρέτηση του της του ε, χρέου και στο πλαίσιο του τη Παγκόσμια Τράπεζα είπε ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση ε, του περίοδου 2017-2020 και υπάρχουν ε, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον οικονομικό ευάλωτο χαρακτήρα τη γεωργία. Καταρχήν, έχει ένα σχετικά μεγάλο ε, εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο. Δεύτερον, που σχετίζεται με αυτό είναι η αύξηση προφανώ των εξωτερικών αποθεμάτων. Και από εκεί και μετά οι απαιτήσει σε ό,τι αφορά το amortization. Άρα λοιπόν ε, παρουσιάστηκε ε, πρόσφατα τον Απρίλιο ε, του 2017 ένα πρόγραμμα που προετοιμάστηκε από κοινού με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως εκτελείται με τον σωστό τρόπο και τον Οκτώβριο του 2017, ε, ε, στο πλαίσιο δηλαδή τη έκθεση που συνέταξε και το προσωπικό από την πλευρά του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, επιβεβαιώθηκε αυτή η σωστή εφαρμογή. Το πρόγραμμα δηλαδή τρέχει με τον σωστό τρόπο, όλοι οι δείκτε απόδοση έχουν επιτευχθεί και βρίσκονται εντό των προβλεπόμενων περιθωρίων, οπότε η σχετική απόφαση από την πλευρά του IMF, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, θα ληφθεί μέσα στο Δεκέμβριο. και με βάση δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που έχει ε, προβλεφθεί, ακριβώ καταδεικνύεται ότι το προσωπικό του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι πολύ ευχαριστημένο με την ε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί τώρα. Το γεγονό ότι ε, το πρόγραμμα θα πρέπει να τρέχει με τον σωστό τρόπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου αποτελεί προπόθεση για την εκταμίευση τη δική μα υποστήριξη και θα υπάρξει ένα μνημόνιο κατανόηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργία που θα περιγράφει τις ε, συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις άσχης της πολιτικής προκειμένου να είναι δυνατόν να ε, λάβει χώρα η εκτέλεση της μακροοικονομικής βοήθειας. Πριν από τρεις εβδομάδες στην Τυφλίδα, στα τέλη δηλαδή Οκτωβρίου, είχαμε προβεί σε μια πρώτη διερευνητικού χαρακτήρα αποστολή στις περιοχές εκείνες που θα μπορούσαν να, να καλυφθούν από το μνημόνιο, εφόσον συμμονηθεί από τους συνομοθέτες, ε, συγκεκριμένα εξετάσαμε τα ζητήματα χρηματοδότησης του δημοσίου και εδώ ε, ειδικότερα την, ε, την σωστή λειτουργία των χρηματικών ροών στην, στην χώρα ακριβώς δικαιούχο τη υποστήριξη, δηλαδή στη Γεωργία, προκειμένου να αποφύγουμε ακριβώ ε, την κατάχρηση αυτών των κονδυλίων και προφανώ ε, η μακροοικονομική υποστήριξη αποτελεί ένα εργαλείο αντιμετώπιση κρίσεων, εξωτερικών δηλαδή κρίσεων, που σημαίνει ότι πρόκειται για μια αρρωγή που δίνεται χωρί πολύ συγκεκριμένε προποθέσει. Δηλαδή δεν είναι μια υποστήριξη που αφορά συγκεκριμένα έργα. Δεν είναι υποστήριξη δηλαδή που θα πρέπει να δαπανηθεί ε, σε κάτι συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά προφανώς η, η χρήση αυτών των κοντιλιών θα πρέπει να γίνεται ε, με νόμιμο τρόπο. Και ακριβώς ε, μία από τις προϋποθέσεις είναι η σωστή εκτέλεση του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της κατάστασης του κράτους. Από εκεί και μετά εξετάσαμε και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις χρηματαγορές, τη χρηματαγορά και το, ειδικότερα το de-dollarization. Ε, παραμένει δηλαδή μία από, ένα από τα τροτά σημεία, αν θέλετε, της ε, οικονομίας της γεωργίας. Από εκεί και μετά ένα τρίτο σημείο ήταν οι κοινωνικές πολιτικές, τις οποίες εξετάζουμε. Ε, η τρέχουσα κυβέρνηση της γεωργίας έχει επιτείνει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να βελτιωθούν τα κοινωνικά συστήματα στη χώρα. Και μία τέτοια λοιπόν προσπάθεια αξίζει τη δική μας υποστήριξη. Για παράδειγμα, επίσης εξετάζουμε την εκπαίδευση, τον τομέα της υγείας, σε ό,τι αφορά δυνητικές δηλαδή αρεσιμότητες εκεί. Και, και ένας τέταρτος ε, τομέας στον οποίο εξετάζουμε είναι ε, το επιχειρηματικό περιβάλλον και η προώθηση ε, των εξαγωγών και, και του εμπορίου. Και εδώ δίνουμε έμφαση στο, στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ε, την SFTA και ε, όπως αναφέρθηκε ήδη από έναν από τους ομιλητέ, προσπαθούμε δηλαδή μέσα στο διαθέσιμο χρόνο που έχουμε να διασφαλίσουμε ότι πράγματι ε, θα δοθεί ο κατάλληλο χρόνο για την εφαρμογή τη. Και είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό εδώ, γιατί προφανώς μια τέτοια συμφωνία της FTA είναι, έχει μεγάλο βάθος χρόνου και η εφαρμογή δηλαδή αφορά ένα πολυετή χρονικό ορίζοντα ενός, ενώ αντιθέτως η μακροοικονομική υποστήριξη είναι ένα εργαλείο αντιμετωπισής κρίσεων και κατά συνέπεια εκταμείωση των σχετικών κοντιλών μπορεί να λάβει η χώρα σε ε, σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από στοιχεία τα οποία ε, βρίσκονται σε φάση προετοιμασία και τα οποία θα μπορούσαν να επιδεχθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη Γεωργία. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση ε, μια νομοθεσία σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει και η οποία εναρμονίζει τις ε, νομικές μορφές που λαμβάνουν επιχειρήσεις, ε, τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων και την εναρμόνιση όλων αυτών των ε, μορφών των εταιριών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα από εκεί και μετά στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης όπως και όλων των άλλων επιχειρήσεων παροχής μακροοικονομικής ε, ε, ενίσχυσης έχουμε και κάποιες ε, πολιτικές ερεσιμότητες. Καταρχήν η διαδικασία της πολιτικής μεταρρύθμισης, κάτι το οποίο ακόμα τρέχει και σχετικά η Επιτροπή της Βενετίας εκπώνησε μια θετική σε γενικές γραμμές έκθεση, οπότε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ε, άποψη τη Επιτροπή αλλά και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θεωρούμε πω εν λόγω αρεσιμότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την πολιτική μεταρρύθμιση πληρείται πράγματι και αυτό αναφέρεται και στην πρόταση από την πλευρά τη ε, Επιτροπή. Επίση αναφέρθηκαν οι δύο προηγούμενε ε, τέτοιε ενισχύσει που έχουν δοθεί στην Γεωργία, η πρώτη το 2008 και η δεύτερη το 2013 που υπογράφηκε δηλαδή το 2013 και ολοκληρώθηκε ε, στις αρχές του 2017. Επειδή ακριβώς ε, ολοκληρώθηκε τόσο πρόσφατα δεν υπάρχει ακόμα μια εξπόσα εκ των υστέρων δηλαδή αξιολόγησή της. πρέπει να παρέλθει δηλαδή κάποιο χρονικό ε, διάστημα από την ολοκλήρωση μιας τέτοια διαδικασίας χρηματοδότησης ε, και την ε, εκπόνηση μιας έκθεσης εκ των υστέρων, γιατί θα πρέπει να συλλέξουμε καταρχήν τα οικονομικά δεδομένα που χρειάζεται να εξετάσουμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν μέσα στο 2018 θα εκπονηθεί αυτή η έκθεση αξιολόγησης για το δεύτερο MFA και θα την εξετάσουμε βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώ θα είναι δημοσία προσβάσιμη, θα δημοσιευτεί δηλαδή και θα μπορείτε όλοι σας ε, και το Συμβούλιο να τη διαβάσει. Αυτές λοιπόν οι των υστέρων αξιολογήσεις αποτελούν μια καλή ευκαιρία για να αναφερόμαστε και στα αποτελέσματα των προηγουμένων λοιπόν ενισχύσεων που έχουν δοθεί και προφανώ θα το πράξουμε και στο μέλλον όπως ανέκαθεν κάνουμε και νομίζω πως την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη συνάντηση θα υπάρξει εδώ ε, ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά συμφωνία MFA εδώ ε, στη συνέντευξη τη ΣΥΝΤΑ. Οπότε θα ε, υπάρξει δυνατότητα να απαντηθούν και περισσότερο ερωτήματά σας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συρρεσιμότητα, τέθηκε ένα συγκεκριμένο ερώτημα από τον Πρόεδρο. Να σας πω λοιπόν ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρόσφατα εξέδωσε γνωμοτήσεις σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις σε σχέση με δύο χώρες, την Ινδονησία και την Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν ε, αυτό το MFA ε, αφορά ένα ολόκληρο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει δηλαδή και άλλες μορφές ενίσχυσης προς αυτές τις δύο χώρες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές και οι δύο αυτές εκθέσεις είναι θετικές και περιλαμβάνουν τόσο επιτεύγματα όσο και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι ερεσιμότητες. και με βάση τα όσα έχει δημοσιεύσει κατά ε, τελευταία χρόνια και πρόσφατα ε, το ελεκτικό συνέδριο δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που σχολεία, όσα σχολιάσατε σε ό,τι αφορά το ε, τις 5 από τις 15 σε ό,τι αφορά λοιπόν το, το, τα ζητήματα του πολιτικού περιβάλλοντος σε αυτές τις χώρες. για παράδειγμα στην Ουκρανία το είδαμε ότι ε, ε, η χρονική περίοδος που κάλυψε ε, η έκθεση αξιολόγηση κάλυψε την περίοδο 2007-2015 και άλλαξαν πάρα πολύ βέβαια σε αυτό το διάστημα και αυτό έχει επιπτώσεις και στην χωρίς της ενίσχυσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις αιρεσιμότητες και τις, σχετικές, τις σχετικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ κλείνοντας για την υποστήριξή σας απέναντι στην πρότασή μας. Ελπίζουμε να λάβουμε την υποστήριξη και της Δικής Επιτροπή και τη ΑΦΕΤ έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην ε, ταχεία έγκρισή της έτσι ώστε να ταμιευτεί ε, ταχύτατα αυτή η υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάκουλα, τον λόγο. Όχι, νομίζω ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα έχουν υποθεί λοιπόν. Ωραία. Τότε θα σας δώσω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 10 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου. 20 Φεβρουαρίου για την Ολομέλεια. Σας περιμένω όλους και πάλι 5 με